Dear colleagues, summer is close and... Αγαπητοί συνάδελφοι, τέλειωσε το καλοκαίρι. Ξαναρχίζουμε τη δουλειά. Ας αρχίσουμε τη συνεδρίασή μας λοιπόν με την υιοθέτηση της ημερήσιας διάταξης εάν δεν υπάρχουν αντιρρήσεις, εγκρίνεται χωρίς τροποποιήσεις. Διερμηνία έχουμε σε 20 γλώσσες σήμερα. Και έχετε σε θέση ηλεκτρονικά το φάκελο για τη συνεδρίαση με τα έγγραφα και βέβαια ξέρετε ότι μεταδίδεται μέσω του διαδικτύου η συνεδρίαση. Έχουμε να επικυρώσουμε πρακτικά τεσσάρων διαφορετικών συνεδριάσεων τις 16-17 Ιουνίου 2015, 8 Ιουνίου 2015, 6 και 7 Μαΐου 2015 και 9 Μαρτίου 2015. Εάν δεν έχετε μέχρι το τέλος της συνεδρίασης εκφράσει αντιρρήσεις, εγκρίνονται τα πρακτικά αυτών των συνεδριάσεων. Συστάσεις των συντονιστών. τις διαθέτουμε ηλεκτρονικά, τις διαβάζετε και αν δεν διατυπηθούν ε, αντιρρήσεις θεωρείτε ότι εγκρίνονται και έτσι περνούμε στην ψηφοφορία. Σας καλώ να χρησιμοποιήσετε την ηλεκτρονική κάρτα. Και ξεκινούμε με τον ε, προϋπολογισμό 2016 και τη σχετική γνωμοδότηση. Παρακαλώ. Πρόεδρε, νομίζω ότι ταλαιπωρήθηκε στι θερινέ διακοπέ η κάρτα μου ηλεκτρονική για τις προφορίε. Γιατί βλέπω ότι δεν δουλεύει πια. Έχω την παλιά μπορώ να τη Είχα και εγώ δυσκολε διακοπέ. Καλά. Λοιπόν, για δοκιμάστε και στη διπλανή σχισμή. Όχι. Δεν δουλεύει τότε θα υπολογίσουμε την ε, ψήφο σας, ε, θα μας επισημαίνετε σε τι θέλετε. Και ξεκινώ με την πρώτη ψηφοφορία, σχέδιο γνωμοδότησης. Και τροπολογία υπαριθμών 1 του κυρίου Καπούτο υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 2 υπέρ κατά αποχές απερίφθη 3 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 4 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 5 υπέρ κατά άποχες εγκρίνεται 6 υπέρ κατά επαληθεύουμε ψήφισαν όλοι πέρας έγκρινεται με μία ψήφο διαφορά Α, καταψηφίζετε εσείς. Απερίφθη λοιπόν. <laughs> Ήταν κρίσιμη η ψήφο σας. Υπαριθμόν 7 υπέρ κατά αποχές εγκρίν. απορρίπτεται 8 υπέρ κατά αποχές επαληθεύουμε. Ψηφίσαν οι πάντες. Εγκρίνεται. 9. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 10. Δύο τμήματα. Πρώτο. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απερίφθη. Δεύτερο υπέρ. Κατά. Αποχές σε Ψηφίσαν οι πάντες πέρα στις ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. 11. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 12. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απερίφθη. 13. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 14 υπέρ. Κατά. Επαλήθευση. Ψήφισαν όλοι πέρα τη ψηφοφορία. Εγκρίνεται. 15. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 16 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται και 17. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Ηλεκτρονικά η τελική ψηφοφορία αρχίζει. Ψήφισαν όλοι. Πέρασε. Έγκρινεται. Και τώρα ψηφοφορίε για τις... λοιπόν, για τον προϋπολογισμό. Ένβη 6113 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 6.114 υπέρ, κατά, αποχές ελέγχουμε. Avete votato tutti? Il voto è chiuso. Ψήφισαν όλοι πέρα στις ψηφοφορίες. Εγκρίνεται. Τώρα. 6.106 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 6.143 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 6.114 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 6.145 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 6.116 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 6.115 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 617 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 618 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 619 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 602 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 604 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 605 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 638 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 607 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 608 υπέρ κατά αποχές ελέγχουμε. Avete votato tutti? Ψηφίσατε όλοι. Πέρας εγκρίνεται. 646 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 641 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 647 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 620 υπέρ κατά εποχές εγκρίνεται 621 υπέρ κατά εγκρίνεται 622 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 640 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 639 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 623 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 648 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 609 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 610 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 611 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 612 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 635 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 636 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 637 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 649 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 124 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 625 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 626 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 629 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 627 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 628 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 631 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 630 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 633 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 6132 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 634 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 6100 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 650 υπέρ κατά αποχές Ελέγχουμε. Ψήφισαν όλοι πέρα τη ψηφοφορία. Εγκρίνεται. 6.101 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Και έτσι ολοκληρώσαμε την ψηφοφορία για τον προϋπολογισμό και σας ευχαριστώ ως συγητής και μπορούμε να πάμε τώρα στο επόμενο σημείο σχετικά με το, με το ατύχημα της ε, κόκκινης σύλληδας στην Ουγγαρία lessons learned κτλ. We start immediately with uh, electronic vote. Πάμε απευθεία στην ηλεκτρονική ψηφοφορία Καταρχά για το θέμα της Επιτροπής. Άρχεται η ψηφοφορία. The vote Πέρας. Εγκρίνεται. Το δεύτερο είναι για το Συμβούλιο επίσης εδώ άρχεται η ψηφοφορία. Everybody at Ψηφίσατε, πέρας, εγκρίνεται. Μάλιστα. Άρα εδώ τελειώσαμε με τις ψηφοφορίες και πάμε στο επόμενο σημείο που είναι η συζήτηση για το αυτό θέμα πέντε χρόνια από το ατύχημα αυτό στην Ουγγαρία και καλούμε όλα τα μέλη που επιθυμούν να αποχωρήσουν να το κάνουν σύντομα αν θέλετε ώστε να συνεχίσουμε την ε, δουλειά μας Έχουμε διάφορους τώρα συνεισηγητές. Θα δώσω όμως ε, το λόγο στον Γιάβορ και μετά θα πάμε στις άλλες πολιτικές ομάδες. Παρακαλώ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω και όλα τα μέλη της Επιτροπής που με υποστήριξαν στη δουλειά αυτή. Ε, στο, στην πέμπτη επέτειο του, του ατυχήματος αυτού καταφέραμε να το βάλουμε στην ε, ημερήσια διάταξη η καταστροφή του Κόλονταρ ήταν από τα μεγαλύτερη κλίμακα σε βιομηχανικά ατυχήματα στην Ουγγαρία με 11 θύματα και πολύ σημαντικές περιβαλλοντικές ε, συνέπειες. Τα συμπεράσματα είναι σε πρώτη φάση για την Ουγγαρία αλλά όχι μόνο. Την στιγμή του ατυχήματος ε, οι ευρωπαϊκοί θεσμοί παρακολούθησαν ε, στενά το θέμα αυτό, την καταστροφή αυτή, διότι υπάρχουν πάρα πολλά εμπειρίες και μαθήματα που μπορούν να είναι χρήσιμα συνολικά για την Ευρώπη και σε ρυθμιστικό επίπεδο, σε νομοθετικό επίπεδο. Πέντε χρόνια αργότερα λοιπόν τοποθετούμε το θέμα στη μέση διάταξη και γιατί είναι χρήσιμο αυτό και απαραίτητο. Και πάρα πολύ σύντομα θα πω το εξής. Προφανώς συνέβησαν διάφορα πράγματα, μεσολάβησαν κάποιες ε, πρόοδοι, ιδιαίτερα για την ε, ουγγρική περιβαλλοντική νομοθεσία, αλλά και εν μέρη και ευρωπαϊκή νομοθεσία. Όμως υπάρχουν και κάποια ερωτήματα που προκύπτουν. Από τη στιγμή που έγιναν οι μελέτες των εμπειρογνωμόνων, υπάρχουν ζητήματα τα οποία δεν έχουν καλυφθεί, δεν έχουν κλείσει και υπάρχουν αρκετές πτυχές ε, σημαντικές ε, και για την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία, δηλαδή περιοχές τις οποίες δεν έγιναν οι πρόοδοι που ελπίζαμε μετά το ατύχημα ότι θα γίνουν. Εάν λοιπόν μια τέτοια καταστροφή, ένα τέτοιο σημαντικό ατύχημα δεν παρκούσε για να σημειωθεί αυτή η πρόοδος, τότε αναρωτιέται κανείς τι πρέπει να γίνει τι περισσότερο πρέπει να γίνει. Άλλη μια τέτοια καταστροφή ώστε να κάνουμε τα βήματα προς τα εμπρός για να αποτρέψουμε τέτοιες περιπτώσεις για το μέλλον. Το πιο σημαντικό συμπέρασμα που μπορεί να εξαχθεί είναι ότι τα συστήματα ελέγχου στην Ουγγαρία δεν ήταν επαρκή πριν το ατύχημα, δεν ήταν σε θέση οι αρχές δεν είχαν τη δυνατότητα να εντοπίσουν τα κρίσιμα στοιχεία που οδήγησαν στο ατύχημα. Εντοπίστηκαν λοιπόν ελλείψεις ή την ανάλυση αντικτύπου που η Κομισιόν θα έπρεπε να έχει υποβάλει και ακόμα δεν την έχουμε δει. Αυτή η ανάλυση περιβαλλοντικού αντικτύπου θα πρέπει να υποβληθεί και δεν μπορεί να είναι μόνο ευθύνη των κρατών μελών. Δηλαδή, ποιο θα πρέπει να είναι το σύστημα περιβαλλοντικού ελέγχου ή επιθεώρησης είναι μια δέσμη, μια πρόταση που πρέπει να φτάσει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, πρέπει να υποβληθεί και αυτό είναι μια ελάχιστη προσδοκία θα έλεγα, ελάχιστη απέτηση. δεύτερο μάθημα που εξάγεται από την καταστροφή του Κολόνταρ όπως είχε συμβεί και στην επιμόλυνση ενός ε, ποταμού το 2010 οι επιχειρήσεις που είναι υπεύθυνε για, ε, για την μόλυνση αυτή, για την περιβαλλοντική αυτή ζημιά, βρίσκουν κενά στις διατάξεις της νομοθεσίας ώστε να μην καταβάλουν τις αποζημιώσεις που πρέπει. Είναι απαραίτητο να έχουμε ένα σύστημα περιβαλλοντικής εξασφάλισης και λογοδοσίας, στην ουσία ευθύνης νομικής, ώστε να ακολουθούμε την αρχή ότι αυτός που επιμολύνει πρέπει να καταβάλει το αντίτιμο, την αποζημίωση το κόστος δηλαδή της αντιμετώπισης της περιβαλλοντικής ε, ζημίας που ακολουθεί. Θα πρέπει να είναι υπεύθυνοι αυτοί που προχωρούν σε αυτές τις μολύνσεις και όχι να αναλαμβάνει όλο αυτό το κόστος και την ευθύνη ο προϋπολογισμός των κρατών μελών και τελικά ο φορολογούμενος πολίτης. Και ακριβώς αυτό συνέβη στο Κόλονταρ. Ε, ε, περί τα 100 εκατομμύρια ευρώ κατεβλήθησαν από το Ουγγρικό κράτος για να αντιμετωπιστεί μια σημεία που προήλθε από μια ιδιωτική επιχείρηση. Έχουμε και ένα άλλο μάθημα που εξάγεται και θα ήθελα να υπογραμμίσω. Δηλαδή αυτό που έχει σχέση με την καλύτερη διαθέσιμη τεχνολογία. Είναι μια έννοια που υφίσταται και μπορεί να χρησιμοποιείται και πρέπει να χρησιμοποιείται σε συγκεκριμένες περιπτώσεις. Στην πράξη όμως δεν χρησιμοποιούμε ε, τις καλύτερες δυνατές λύσεις υπό την περιβαλλοντική και επιστημονική τεχνική έννοια. Από πλευρά δηλαδή των επιχειρήσεων. Είναι λοιπόν απαραίτητο να εξετάσουμε την πρακτική ή στην εφαρμογή, στην τήρηση της έννοιας αυτής, ώστε η ευρωπαϊκή βιομηχανία να χρησιμοποιεί τις καλύτερες διαθέσιμες τεχνολογίες μεθόδους ώστε να αποτρέπεται κρούσμα αντίστοιχου ατυχήματος, αντίστοιχης ε, καταστροφής όπως αυτό που συνέβη στην Ουγγαρία. Δεν είναι, επαναλαμβάνω, πρόβλημα των μεμονωμένων κρατών μελών. Είναι θέμα των ευρωπαϊκών θεσμών, της Κομισιόν και του Κοινοβουλίου του συνολό του, θα έλεγα. Εγώ θα ήθελα να ευχαριστήσω όλου του συναδέλφους που ζήτησαν να τοποθετηθεί το θέμα αυτό στην ημερήσια διάταξη. Και νομίζω ότι μπορούμε και την Εκτελεστική Επιτροπή μπορούμε να υποβάλουμε ένα ερώτημα και περιμένουμε από την Εκτελεστική Επιτροπή ένα, μια ικανοποιητική και πλήρη απάντηση απέναντι στα προβλήματα που έχουν σημειωθεί. Ευχαριστούμε Γιάβο να δώσω το λόγο τώρα στους υπόλοιπους συνεισηγητές ο κύριος Χολβενή Ευχαριστώ πολύ Είχαμε ένα ε, μάθημα Ουγγρικών μεγάλη ευκαιρία οπότε και εγώ θα συνεχίσω στα Ουγγρικά που είναι επίσης η μητρική μου γλώσσα γιατί δεν έχουμε πάντοτε τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσουμε ε, τα Ουγγρικά. Πρώτα απ' όλα λοιπόν, ήθελα να ευχαριστήσω. Πρώτα απ' όλα θέλω να ευχαριστήσω τον κύριο Γιάβορ για το υλικό που μας διένυμε. Είναι νομίζω σωστή η προσέγγιση. Το πρόβλημα είναι σημαντικό. Πρέπει οπωσδήποτε να το συζητήσουμε, να το αντιμετωπίσουμε. Και δεν νομίζω ότι θα προξενούσε, θα οδηγούσε σε περαιτέρω επιθέσεις βάρο τη Ουγγαρία σε ένα τέτοιο πρόβλημα, όπω είδαμε τις τελευταίες εβδομάδε. γιατί πρόκειται για πρόβλημα διαφορετική φύσεω. Είναι ένα ζήτημα που αφορά όλη την Ευρώπη και βεβαίως θα πρέπει να διερευνήσουμε πού βρίσκονται οι αδυναμίες σε επίπεδο Ουγγαρίας, πού είναι τα κενά. Αλλά βέβαια δεν χρειάζεται να γίνεται κριτική όπου δεν είναι αυτή αναγκαία. Η Ερυθρά Ηλής έχει πάρει μια σημασία ως έκφραση στα ουγγρικά για πολλές περιοχές του Ουγγαρίας Έχουμε εντωμεταξύ 11 νεκρούς από την καταστροφή αυτή και πολλοί άριθμους τραυματίες. Η καταστροφή βρήκε απροετοίμαστε στις υπηρεσίες του Ουγγρικού κράτους και νομίζω ότι μετατρέπεται και όλα σε ένα εμβληματικό ατύχημα αυτό Πολλά είναι αντίστοιχα, πολλά είναι τα αντίστοιχα ατυχήματα που έχουν λάβει χώρα, αλλά με αυτό ιδιαίτερα καταδεικνύονται οι διαστάσεις του προβλήματος, όπως είπε και ο συνάδελφος νωρίτερα. Γι' αυτό νομίζω ότι πρέπει να το συζητήσουμε. Δεν μπορεί εδώ να υλοποιηθεί η αρχή του ρηπαίνων πληρώνει. Μιλούμε για εκατομμύρια, εκατοντάδες εκατομμύρια επιβάρυνση για το ουγγρικό κράτος επειδή η επιχείρηση που προξένησε την φυσική αυτή καταστροφή ήταν ε, σε πτώχευση, πτώχευση του μεταξύ. Δεν ικανοποιούνται λοιπόν οι όροι του ορυπαίνων πληρώνει. Το οποίο πρέπει να ισχύει, αλλά στην πράξη οι επιχειρήσεις δεν έχουν προβλέψει κονδύλια για την κάλυψη των αποζημιώσεων για τις ζημίες που έχουν προξενήσει είτε στην ίδια την Ουγγαρία είτε στην ευρύτερη Ευρώπη. Και έτσι δεν τηρούνται οι όροι του πέραν πληρώνει και καλούνται το δημόσιο να καλύψει αυτή την ζημιά. Και έτσι θεωρητικά θα μπορούσαν να έχουν στα θέση τους εναλλακτικέ πηγές ε, χρηματοδότησης των αποζημιώσεων. Είναι μάλιστα το ζήτημα αυτό το οποίο είχε υπογραμμίσει ο Επίτροπος για το περιβάλλον την εποχή ο Κίνη και ο κύριος Γιάννος είχε επιμείνει ιδιαιτέρως στο ότι δεν υπήρχαν επαρκείς πόροι και ότι δεν θα υπήρχαν επαρκείς πόροι σε περίπτωση ατυχήματος. Είναι λοιπόν απαραίτητο να συνεργαστούμε εμείς τα θέματα αυτά, με έμφαση ιδιαίτερα της υποχρέωσης για αποζημίωση του ρηπαίνοντα. Και μπορούμε να αντλήσουμε και άλλο δίδαγμα από την καταστροφή αυτή. γιατί θα χρειαστεί να συζητήσουμε και απόβλητα ορυχείων, ένα καυτό ζήτημα. Θα το συζητήσουμε και αυτό εν συντομία. Είναι πολύ σημαντικό όμως με τη συζήτηση αυτή να μην επαναλαμβάνουμε τα ίδια επιχειρήματα. Γιατί είναι στο ευρύτερο πλαίσιο η προβληματική η ίδια. Άρα λοιπόν, καλό θα ήταν να μην επαναλαμβάνουμε τα ίδια λόγια. Όπως είπα υπάρχουν δύο σημεία του κυρίου Γιάρο και θέλω και εγώ να υπογραμμίσω και το ζήτημα της ασφάλισης ή της πρόληψης, της πρόβλεψης ε, ικανοποιητικής αποζημίωσης. Ξέρουμε ότι θα έχουμε την ευκαιρία πάλι τον Ιανουάριο δε να συζητήσουμε τα θέματα αυτά, γιατί όπως είπα, η... Ε, το πρόβλημα αφορά όχι μόνο την Ουγγαρία αλλά και τα άλλα κράτη-μέλη και δεν χρειάζεται μόνο να υπάρχουν διδασκαλίες και διδάσκοντες, αλλά και μαθητές και μαθητευόμενοι. Ευχαριστώ πολύ, Ζάνη. Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Πρόεδρε, Υπήρξε μια πολύ εντατική παροπαρασκευαστική ε, διαδικασία πριν από το καλοκαίρι και θα ήθελα να σας ευχαριστήσω όλους για τη συμμετοχή σας. Εμείς ε, ως ε, σοσιαλδημοκράτες ε, είμαστε ικανοποιημένοι με το περιεχόμενο της προφορικής ερώτησης, όπως επίσης και με την κύρια, πρόταση, με την κύρια πρόθεση της ε, πρότασης ε, ψηφίσματος. Σαφώς υπάρχει κοινή κατανόηση του γεγονότος ότι πρέπει να γίνουν κάποια βήματα για την περιβαλλοντική πτυχή, το τονίζω αυτό, της εξορυκτικής, της πιο συστηματικά. Θα πρέπει να καλέσουμε επιγόντως την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να ε, κάνει ε, βήματα προς την εφαρμογή της ενωσιακής νομοθεσίας ε, ως προς τις επιθεωρήσεις για να δούμε τι διδάγματα έχουμε από την καταστροφή αυτή της ερυθράς ηλίως όπως επίσης και να υπάρξουν επαρκείς οικονομικοί μηχανισμοί για την ενίσχυση του περιορισμού της καταστροφής μετά ε, την ε, ε, καταστροφή. Εννοώ να υπάρξουν, πρέπει να υπάρξουν και κλείνει το μικρόφωνο του Μιλική. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να μην υπάρχουν υποκειμερικοί υποκειμενικά στοιχεία, ε, να μην υπάρξουν ε, ε, έπαινοι για συγκεκριμένες κυβερνήσεις ή συγκεκριμένες επιχειρήσεις. Δεν είναι τώρα το κατάλληλο, η κατάλληλη στιγμή ούτε το κατάλληλο έγγραφο για να κάνουμε πολιτικές ανακοινώσεις. Το σημαντικό είναι η προστασία του περιβάλλοντος. Ε, κάτι το οποίο υπόθηκε και στο παρελθόν, θα μπορούσα να συνεχίσω να το τονίζω, η σημασία της οικονομικής διαφάνειας ε, των ε, ταμείων περιβαλλοντικής αποκατάστασης, όπως επίσης και η συμμετοχή της κοινωνίας των πολιτών σε τέτοιου είδους περιπτώσεις. Δεν έχουμε τελειώσει τη δουλειά μας, κύριε Πρόεδρε, οπότε θα ήθελα να καλέσω όλους σας να συνεχίσουμε να συμμετέχουμε σε αυτή την προσπάθεια για να επιτύχουμε όσο το δυνατόν καλύτερα αποτελέσματα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ και εγώ. Δεν έχουμε εκπρόσωπο της ECR. Δεν ξέρω αν η Γκου εκπροσωπείται και θέλει να λάβει το λόγο. Έχετε το λόγο. Η κυρία Κονέτσνα δεν είναι εδώ η συνάδελφός μου, ε, οπότε την εκπροσωπώ. Θα ήθελα καταρχάς ε, να ε, πω συλληπιτήρια στις οικογένειες όλων των θυμάτων, των θυμάτων αυτής της φρικτής καταστροφής στην Ουγγαρία πριν από πέντε χρόνια. Αυτό το ε, ατύχημα ε, έχει δείξει, όπως και άλλα ατυχήματα τέτοιου είδους, ε, ή τέτοιου είδους δείχνουν ότι πρέπει τα απόβλητα της εξοριστικής βιομηχανίας να την χάνουν καλύτερης διαχείρισης. Η εφαρμογή της ενωσιακής, σχετικής ενωσιακής νομοθεσίας είναι πάρα πολύ σημαντική. Πρέπει να υπάρξει και βελτίωση της υφιστάμενης νομοθεσίας για την προστασία της ανθρώπινης υγείας και του περιβάλλοντος. Επίσης θα θέλαμε να δούμε καλύτερο έλεγχο και ενισχυμένη επιθεώρηση ε, των ε, υπαρχόντων ε, ε ορυχείων να υπάρξει καλύτερη προστασία της ανθρώπινης υγείας και του περιβάλλοντος μέσω της βελτίωσης της τρέχουσας νομοθεσίας. Επίσης ζητούμε καλύτερη εφαρμογή της νομοθεσίας ε, δηλαδή να μην ξεχνούμε την κοινωνική ευθύνη των ε, επιχειρήσεων ε, που προβαίνουν και εκμεταλλεύονται την εξορρυκτική δραστηριότητα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο κύριος Φετισίνη. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Εγώ συμφωνώ και προσυπογράφω απολύτως τα όσα είπε ο συνάδελφος Γιάβορ. Πρέπει να εξαγάγουμε διδάγματα από τέτοια κρούσματα γιατί έχουμε ξεκάθαρη ευθύνη εδώ για, τα, για τους ε, ευρωπαϊκούς θεσμούς ε, που δεν είχαν κατανοήσει προηγουμένως ε, πόσο επικίνδυνες είναι αυτές οι περιπτώσεις της, του χειρισμού της κόκκινης ηλίως. Αλλά πρέπει να καταλάβουμε πώς μπορούμε να αποτρέπουμε τέτοιου είδους κρούσματα και αντίστοιχα κρούσματα, αντίστοιχα ατυχήματα. Τι μπορούμε λοιπόν να διδαχθούμε. Καταρχά, κατά την άποψή μας πρέπει να προσέξουμε αυτά που μας λένε οι πολίτες. Γιατί πολλοί πολίτες καταγγέλουν αντίστοιχες και χειρότερες ακόμα ελλείψεις από αυτές. Μετά εδώ έρχονται κάποια μέλη, κάποιοι βουλευτές, τα παρουσιάζουν αυτά στο Κοινοβούλιο, τα παρουσιάζουν στις αρμόδιες επιτροπές, δεν γίνεται τίποτα όμως. Και πολλοί συνάδελφοι της ομάδας έχουν μιλήσει επανειλημμένως για ανάλογες περιπτώσεις πολύ πιο σοβαρές ε, όπως με αυτή της Ουγγαρίας, ιδιαίτερα στη Σαρδινία στην Ιταλία, αλλά δεν έχει γίνει τίποτα. Εκατοντάδες άνθρωποι χάνουν τη ζωή τους από κάθε είδους ρήπων στην Terra dei αλλά δεν συμβαίνει τίποτα. Έχουμε πλήρη αδυναμία να αντιδράσουμε, να αντιμετωπίσουμε αυτά τα θέματα και αυτοί που καταβάλουν το κόστος με διάφορους τρόπους είναι οι πολίτες. Είναι ακάλυπτοι σε ρήπους, σε μόλυνση, δεν προστατεύεται η υγεία τους και από τη στιγμή που δεν παρεμβαίνει με μια οικονομική ενίσχυση η Ευρωπαϊκή Ένωση, καταβάλουν και το κόστος Τη οποιασδήποτε αντιμετώπιση, αποζημίωση κτλ. Και καταβάλουν και το κόστος του προστίμου όταν έρχεται μετά η Ευρωπαϊκή Ένωση και επιβάλλει πρόστιμο παραβίασης ή παράβασης. Επομένως η αρχή ορυπαίνων πληρώνει θα πρέπει να επιβάλλεται. Και με ποιο τρόπο θα επιβάλλεται με αδειοδότηση που θα πρέπει να παρέχεται μόνον όταν υπάρχει οικονομική εγγύηση της δραστηριότητα που διεξάγεται. Σε περίπτωση δηλαδή ατυχήματο. Αλλά αυτό δεν συμβαίνει. Το βλέπουμε χιλιάδες φορές στο πεδίο, στις ε, χώρες μας, στις πόλεις μας, στις περιφέρειές μας. Η αδειοδότηση γίνεται από πολιτικούς που ποτέ δεν καταβάλουν κανένα τίμημα και κανένα κόστος σε επιχειρήσεις που δεν έχουν απλούστατα τη δυνατότητα να αντιμετωπίσουν, να αναλάβουν το κόστος και την ευθύνη τέτοιων τραγικών επεισοδίων. Σας ευχαριστώ κύριος Μπάλτσο. Ευχαριστώ πολύ για τη λόγο που μου δίνετε κύριε Πρόεδρε. Και τη δίνουμε μέλος επιτροπής. Θα να κάνω μια προσωπική ε, παρατήρηση. Την ώρα που ξέσπασε αυτή η καταστροφή, συνεδρίαζε το Ουγγρικό Κοινοβούλιο και μέλη της πολιτικής μας ομάδας αποχώρησαν αμέσως για να πάνε στην περιοχή και να διαπιστώσουν η διεισόμαση το μέγεθος της καταστροφής. Αυτά που σας λέω λοιπόν τώρα στηρίζονται στις προτάσεις του τότε Προέδρου της Επιτροπής του Περιβάλλοντος. Είναι θλιβερό το ότι πέντε χρόνια μετά την καταστροφή αυτή έχουμε ακόμα την υποχρέωση να διατυπώνουμε ερωτήσεις προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή προκειμένου να την ενθαρρύνουμε να αναλάβει νομοθετική πρωτοβουλία για τα θέματα αυτά ή μέτρα για την αποτροπή των καταστροφών. Και είμαστε πολύ επιφυλακτικοί για την επιτυχία αυτών των διαθυμάτων κοινοβουλευτική μα επιτροπή ήταν η μόνη η οποία μέχρι τώρα είχε επιδείξει αίσθημα ευθύνη στο επίπεδο κοινοβουλευτική ε, Ουγγαρία. Ε, η δικαιοσύνη έκανε ό,τι μπορούσε από πλευρά τη μεν, αλλά λίγα κατάφερε μέχρι τώρα. Τουλάχιστον σε πρώτο βαθμό. Και παραμένουν ακόμη πολλές λεκάνες αυτής της ερυθράς ηλίως που παραμένουν επικίνδυνες και τι είχε υποσχεθεί ότι δεν θα επαναλαμβανόταν ποτέ τέτοια καταστροφή ο, καταστροφή ο υπουργό. Είναι ιδιαίτερα επικίνδυνη αυτή η ερυθραηλής, τοξική, μπορεί να προξενήσει δερματικά προβλήματα και πρέπει να ξεπλένεται αμέσως μετά την επαφή με το δέρμα, με την επιδερμίδα, ε, για να αποφευθούν ε, οι συνέπειες της. Εν τω μεταξύ όμως πρέπει να προχωρήσουμε σε μια λύση σε σχέση με τις αποζημιώσεις, οι οποίες δεν πρέπει να καταβάλλονται από τον εθνικό προϋπολογισμό. Και ένα άλλο ζήτημα που θέλω να θίξω έχει να κάνει όχι με τα μεγέθη που μπορεί να προκύψουν τέτοια καταστροφή, αλλά με αυτόν τον ληστρικό καπιταλισμό που επικράτησε μετά την πτώση του ε, και την ε, διάλυση Σοβιετικής Ένωσης και την συμπεριφορά αυτών των ε, επιχειρήσεων που οδηγούν σε τόσα προβλήματα για τους πολίτες. Κοινωνικοί παράγοντες λοιπόν θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη και οι επιχειρήσεις και τα διευθυντικά του τελέχη θα πρέπει να ε, διώκονται και να ε, προσάγονται στη δικαιοσύνη. Ευχαριστώ τον Νάρο. Τον Άνω. Ευχαριστώ πολύ. Η καταστροφή της Ερυθράς Ηλίως ε, αφορά δύο πτυχές που πρέπει να λάβουμε υπόψη. Πρώτον, ο χαρακτήρας ε, ε, μιας βιομηχανίας που λειτουργεί σε μελαμφασμένο τρόπο και ευθύνεται εάν η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να αλλάξει την νομοθεσία πρέπει να το κάνει ενισχύοντας τις απαιτήσεις ασφαλείας. Οι δεξαμενές αποθήκευσης πρέπει πρέπει να έχουν ε, ένα βιβλίο πορείας ε, πολύ πιο αυστηρό και πρέπει και ε, σε ευρωπαϊκό και σε εθνικό επίπεδο να υπάρξει ένα πρωτόκολλο ενημερωμένο. Πρέπει να λάβουμε υπόψη μια δεύτερη διάσταση που είναι η χωροταξία και τα, η, η τοπική ο τοπικός εξοπλισμός, η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν μπορεί να απαντάει σε όλα τα προβλήματα που υπάρχουν σε τοπικό επίπεδο και δεν είναι δυνατόν να υπάρχουν μόνο ευρωπαϊκές ρυθμίσεις. Ε, ε, ε, υπάρχουν βέβαια συστάσεις σε σχέση με, τις τοπικές, με τους τοπικούς μηχανισμούς πρόληψης, όμως η Ένωση δεν μπορεί να παρεμβαίνει σε τοπικού χαρακτήρα προβλήματα. Πρέπει να ενημερώνει τους πολίτες Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά και τις τοπικές αρχές επιστήσω την προσοχή και το, προ, το πρόβλημα ορισμένων εγκαταστάσεων ε, βιομηχανικού χαρακτήρα σε, κάποια κράτη-μέλη. Ο εξυγχρονισμός τους είναι πάρα πολύ σημαντικός, αλλά το κόστος είναι πάρα πολύ υψηλό. Ε, θα ήταν καλύτερο να υπάρξει στόχευση ε, των ταμείων εγγυήσεων για σχέδια αναδόμησης, ανασυγκρότησης, σε, ειδικότερα σε χώρους κοντά στις αστικές περιοχές, κάτι το οποίο θα ήταν πολύ σημαντικό ο όφελος ε, ε, έναντι της, ε, του, του απλού βιομηχανικού κέρδους. Ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Πρόεδρε και ευχαριστώ πάρα πολύ λέει η κυρία Ριβασή για, τον, για το, το, το, τον εισηγητή για το θέμα που έθεσε. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να ε, λάβουμε υπόψη αυτά τα διδάγματα από την καταστροφή αυτή. Δύο πράγματα. Πρώτον, και το είπατε όλοι οι συνάδελφοι, υπάρχει η κοινωνική και περιβαλλοντική ευθύνη των, ε, των επιχειρήσεων, η ενίσχυση των επιθεωρήσεων, η αρχή ρηπαίνων, πληρώνει και οι αδειοδοτήσεις, ε, όπω επίση και το θέμα ε, της φερεγγιότητας των επιχειρήσεων. Αν κάποια επιχείρηση πτωχεύσει, ποιο πληρώνει. Συχνά οι φορολογούμενοι τη χώρα πληρώνουν. Πρέπει λοιπόν να υπάρξουν εγγυήσεις ε, ώστε να ε, ξέρουμε ποιος πληρώνει στην περίπτωση της καταστροφής. Υπάρχουν όμως γενή προβλήματα και είναι το θέμα της διαδικασίας στη Γαλλία. Έχουμε ένα εργοστάσιο το οποίο εξορίζει αλουμίνιο βάση από το βοξίτη και το μεγάλο πρόβλημα είναι αυτή η ερυθρά το, το σύστημα της Ουγγαρίας είναι να συγκεντρώνει όλα αυτά τα παραπροϊόντα σε συγκεκριμένες δεξαμενές, αλλά δεν είναι μόνο τα... υπάρχουν και τα βαρέα μέταλλα, δεν υπάρχουν μόνο τα... Ε, οι τοξικές ουσίες, ε, ε, η ερυθρά υλής. Τι κάνουμε στην, στη Γαλλία, ε, σε 57 χιλιόμετρα έχουμε ε, κάνει μια, έναν τρόπο διοχέτευση όλων αυτών των αποβλήτων στην Μεσόγειο θάλασσα. υπάρχει όμως ένα πρόβλημα σε επίπεδο αυτών των αποβλήτων μήπως πρέπει να υπάρξει μια οικονομική ενίσχυση και εδώ η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει ένα ρόλο να διαδραματίσει πώς θα μπορούσαμε να έχουμε μια κυκλική οικονομία γιατί αυτά τα απόβλητα ε, είτε πηγαίνουν σε μία δεξαμενή. Αν υπάρχει ένας πραγματικός έλεγχος στο σημείο εξόριξης, ίσως είναι μία λύση. Αλλά άμα τα θέλουμε στη Μεσόγειο θάλασσα, ε, τότε όλο το οικοσύστημα και υπάρχουν πάρα πολλές μελέτες αυτή τη στιγμή από ε, την Υπουργό Οικολογίας που λέει ότι υπάρχουν ε, ε συνέπειες για την αναπαραγωγή των ηχθείων κλπ. Το θέμα λοιπόν της διαδικασίας της βιομηχανικής είναι πρόβλημα. Πρέπει να υπάρξει μια συμβατότητα με τη ζωή και την ασφάλεια και την υγεία, ε, διαφορετικά θα πρέπει οι επιχειρήσεις να βρουν μια διαφορετική λύση σε σχέση με τα απόβλητα αυτά. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο κύριος Νάκη. thank you. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Αν μου επιτρέπετε, θα μιλήσω και εγώ στα Ουγγρικά, παρότι στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εκπροσωπώ τη Σλοβακία. Σε αυτήν ακριβώς την ε, περίοδο ήμουν υπεύθυνο ε, του Υπουργείου Περιβάλλοντος ε, στη Σλοβακία, στην περίοδο δηλαδή του ατυχήματος και καθότι είναι ε, η γειτονική μας χώρα η Ουγγαρία το ατύχημα αυτό είχε επηρεάσει και τη δική μας χώρα. Έχουμε και τα ύδατα του Δουνάβεως τα οποία διατρέχουν και τη δική μας χώρα και πρέπει πράγματι να καλύψουμε τα κενά που έχουμε για να μπορέσουμε να αποτρέψουμε τέτοια ατυχήματα για το μέλλον. Υπάρχουν λοιπόν διασυνοριακές διαστάσεις των ατυχημάτων και των καταστροφών αυτών και συμφωνώ ότι δεν μπορούν αυτές οι συνέπειες να περιορίζονται και οι ευθύνες να υφίστανται μόνο για τα κράτη-μέλη. Υπάρχει μια διάσταση χρηματοδοτικής ε, κάλυψης ε, των επιχειρήσεων, των ιδιωτικών, αλλά πολύ συχνά μετακυλίονται όλα αυτά ή στους προϋπολογισμούς των κρατών μελών και μάλιστα των μικρών κρατών μελών. Εξ ονόματος λοιπόν ε, της ε, Σλοβακικής κυβέρνησης μαζί με τους ε, τέσσερις του Βίτσεγκραντ την εποχή εκείνη είχα υποβάλει μια πρόταση στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο ώστε να δημιουργηθεί ένα κοινό ασφαλιστικό ταμείο ένα ταμείο ασφάλισης έναντι καταστροφών είχε προκύψει μια προφορική υπόσχεση δέσμευση η συνέχεια άγνωστη, τουλάχιστον σε εμένα. Δηλαδή ένα ταμείο που θα μπορούσε να είναι μια, ένα ταμείο αλληλεγγύης αν θέλετε. Κάτι τέτοιο υπάρχει, έχει ήδη ε, δημιουργηθεί στις Ηνωμένες Πολιτείες, ένα super fund όπως το ονομάζουν, που είναι πολύ αποτελεσματικό για ευρεία κλίμακα σε βιομηχανικά ατυχήματα. Και εδώ θα έπρεπε να τονίσουμε και μια άλλη πτυχή. Ένα τέτοιο ταμείο θα μπορούσε να είναι πάρα πολύ χρήσιμο για να αντιμετωπίσουμε καταστροφές, ε, βιομηχανικές καταστροφές του παρελθόντος που συνεχίζουν να έχουν συνέπειες. Εάν καταφέρναμε τελικά να έχουμε ένα ταμείο ασφάλισης κοινό που να καλύπτει ακριβώς τέτοιου είδους δαπάνες μια τέτοια οργανωτική δομή αντιστοίχως προς τα όσα συμβαίνουν και στις Ηνωμένε Πολιτείες, θα μπορούσε να αναλαμβάνει και ένα ρόλο ελέγχων και επιθεωρήσεων διότι προκειμένου να επιβάλλουμε την υλοποίηση της αρχής ορυπαίνων πληρώνει, θα πρέπει να έχουμε ελέγχου. Και παράλληλα θα πρέπει αυτό να μην είναι αποτρεπτικό και ε, εξαιρετικά αρνητικό για τον βιομηχανικό κλάδο. Δεν θα πρέπει δηλαδή να μειώνει την ανταγωνιστικότητα συνολικά του κλάδου. Επομένως ένα κοινό ταμείο θα είχε περισσότερο τη δυνατότητα να το αναλαμβάνει αυτό και να επιμερίζει αν θέλετε πιο ισότιμα την ευθύνη. Εγώ θα πρότεινα να υποβάλουμε εκ νέου μια τέτοια πρόταση στην Κομισιόν. Σας ευχαριστώ. Ας ακούσουμε τώρα και την Κομισιόν για το σχέδιο αυτό ψηφίσματος. Θα δώσω το λόγο στον εκπρόσωπο της Κομισιόν. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Η Επιτροπή θα ήθελα να ευχαριστήσει το Κοινοβούλιο για το ενδιαφέρον που επιδεικνύει εν γέννη για τα περιβαλλοντικά ζητήματα και ιδιαίτερα που επιτρέψει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή να αναλογίσει τα διδάγματα που προκύπτουν από το δυστύχημα που έλαβε χώρα πριν από πέντε χρόνια. Βεβαίω η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα προσφέρει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο κάθε δυνατή πληροφορία έχουμε συλλέξει για το δυστύχημα τις συνέπειες του και τις δράσεις που ανελήφθησαν από όλους τους εμπλεκόμενους φορείς. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ιδιαίτερα θα δώσει σημασία στην αξιολόγηση την οποία ζητεί η πρόταση ψηφίσματος, ε, όταν υιοθετηθεί βεβαίως ε, από το Κοινοβούλιο, και θα αξιολογήσει τη δυνατότητα για παρακολούθηση ονδήποτε επιμέρους ε, προτάσεων εξετάζει ενδεχομένως το Κοινοβούλιο. Όπως και να έχει η Επιτροπή αναμένει από το Κοινοβούλιο με τις πολλές του ερωτήσεις και τις ακροάσεις του ε, να δει ότι και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει ε, υλοποιήσει πλήρως τις ε, διατάξεις και τα μέτρα εκείνα τα οποία επιτρέπουν την αποτροπή ή ελαχιστοποίηση συνεπειών ε, τέτοιου είδου ατυχημάτων. Σε κάθε περίπτωση όμως η ευθύνη για την υλοποίηση των μέτρων αυτών ε, ανοίξει τα κράτη-μέλη. Του του λεχθέντος ενδέχεται σε ορισμένε περιπτώσεις η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να εξετάσει τον ενδεχόμενο βελτίωση των νομοθετημάτων, όπω άλλωστε ζήτησαν ορισμένοι από του ευρωβουλευτέ που τοποθετήθηκαν νωρίτερα. Πριν όμω κατατεθεί οποιαδήποτε νέα τέτοια πρόταση ή μέτρο, θα πρέπει να εκτιμηθεί εάν το ισχύον πλαίσιο υλοποιείται επαρκώ και αν αποδίδει όπως αναμένεται. Όπως και να έχει, ευχαριστώ Πρόεδρε και περιμένουμε με ενδιαφέρον να διαβάσουμε το τελικό κείμενο για την ε, πρόταση ψηφίσματος. Ευχαριστώ πολύ λίγο Πρόεδρος και πριν κλείσουμε το θέμα αυτό της ημερήσιας διάταξης θα πρέπει να σας υπενθυμίσω το χρονοδιάγραμμα. Τροπολογίες μπορούν να κατευθούν έως τις 6 το απόγευμα σήμερα ψηφοφορία στην Επιτροπή μας στις 22 Σεπτεμβρίου, στη Δε Ολομέλεια, στην πρώτη Ολομέλεια του Οκτωβρίου. Και έτσι περνώ στο προσοχές μας θέμα, στο επόμενο θέμα, που είναι ανταλλαγή απόψεων ε, με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, την Προεδρία του Συμβουλίου, για την ε, διαδικασία επαλήθευσης σε πραγματικές συνθήκες οδήγησης ε, για οχήματα ελαφρά και δίνω το λόγο ξεκινώντας στην Επιτροπή προκειμένου να μας εκθέσει τις επόψεις της Επιτροπής για τη διαδικασία επαλήθευσης σε όρους πραγματικής οδήγησης η κυρία Σίσκο φυσικά, εκ μέρους Ευρωπαϊκής έχει το λόγο. Ευχαριστώ. Πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ. κύριε και κύριοι, καλημέρα σα. Θα ήθελα να σα ευχαριστήσω για την ευκαιρία που μας προσφέρετε να σας εκθέσουμε τις εξελίξεις και τη δουλειά μας σε σχέση με το πακέτο αυτό. Θα χρησιμοποιήσω μια παρουσίαση σε PowerPoint ε, για να σας εξηγήσω τα θέματα που έχουμε. Θα δείτε ποια είναι τα πραγματικά αισθήματα που αντιμετωπίζουμε και ενδεχομένως να ένα σκοπό νωρίτερα να δώσω κάποιες πληροφορίες σε σχέση με την εξέλιξη των συζητήσεων, προκειμένου να δώσω κάποιε πληροφορίε σε σχέση με την εξέλιξη των συζητήσεων στην Επιτροπή, θα ήταν καλό να σα δώσω κάποιε πληροφορίε για την έκταση του προβλήματο και να δώσω το υπόβαθρο όλη αυτή τη ε, πρόταση. Γιατί λοιπόν έχουμε το, η πρόταση αυτή, πώ θέλουμε να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα και στη συνέχεια θα σα πω που βρισκόμαστε και τι σκοπεύουμε να κάνουμε τι επόμενε εβδομάδε και μήνε. Ο λόγο για τον οποίο συζητούμε το RDE τις πραγματικές ε, εκπομπές ε, συνθήκες οδήγησης έχει να κάνει με την ε, προστασία του περιβάλλοντος και την υπέρβαση ορίων εκπομπών ιδιαίτερα εξαρτικά κέντρα από τα κράτη-μέλη. Ο κύριος λόγος για τον οποίο να αντιμετωπίσουμε την κατάσταση αυτή προέρχεται κατά βάσα πιθανότητα από εκπομπές οχημάτων που χρησιμοποιούν βενζίνη, δίζελ, πετρέλαιο δίζελ και διαπιστώνουμε ότι σε 20 κράτη-μέλη υπάρχει υπέρβαση των ορίων, ε, κατά των οποίων των μελών μάλιστα έχουμε κινήσει διαδικασίες η Αυτό δείχνει πόσο σοβαρό είναι το πρόβλημα. Είμαστε βέβαια υποχρεωμένοι να συνεχίσουμε να επιταχύνουμε και να ολοκληρώσουμε τη δουλειά μας για τις πραγματικές εκπομπές συνθήκες οδήγησης, το ταχύτερο δυνατό. Υπάρχουν διμερεί ε, όρια για τα ε, οξύδια του αζότου. Τα έχουμε παρακολουθήσει και αντίστοιχα προσαρμόζουμε την νομοθεσία. Θα ήθελα να επενθυμίσω ότι την πρώτη, από την 1η Σεπτεμβρίου μπαίνουν, ε, τίθεται σε ισχύ για όλα τα καταχωρημένα αυτοκίνητα οι προϋποθέσεις και τα όρια για το επίπεδο Ευρώπης, των, ε, Ευρώπης 6. Αλλά βέβαια θα πρέπει να παρακολουθούμε και τι συμβαίνει στην πραγματικότητα. Αυτός άλλωστε είναι και ο πυρήνας του προβλήματος. Και αυτό είναι το ζήτημα το οποίο πρέπει να αντιμετωπίσουμε το κενό μεταξύ των πραγματικών συνθήκων οδήγησης και των εκπομπών τους και των δοκιμών οδήγησης κυρίως εντοπίζεται στα οξύδια του αζότου. Θα δούμε και άλλα ρηπαντές αργότερα, αλλά αυτή τη στιγμή επικεντρωνόμαστε στα οξύδια του αζότου. Θα θυμάστε ίσως ότι είχαμε ε, θεσπίσει μια ομάδα εργασία το 2011 συγκεκριμένα για να παρακολουθήσει αυτέ τι διαδικασίε και να, δει, να βρει διαδικασίε δοκιμών που θα μπορούσαν να επαληθεύσουν πραγματικέ συνθήκε οδήγηση και τι εκπομπέ του. Έχει προχωρήσει αυτή η δουλειά και έτσι έχουμε φτάσει στην έννοια του RDEs που είναι οι πραγματικέ εκπομπέ οδήγηση. Μια πρόταση που δεν είναι άλλωστε καινούρια, γιατί ήδη είχαμε στις προτάσεις του Euro 5 και του Euro 6, επίπεδο 5 και 6, ε, δώσει αντίστοιχε παραπομπέ. Δύο στοιχεία είναι σημαντικά για, το, για την όλη δέσμη μέτρων. Πρώτον, ο τρόπος με τον οποίο θα γίνονται οι εκπομπές σε πραγματικές συνθήκες, στην πραγματικότητα και αυτό είναι και ο λόγος για τον οποίο έχουμε θεσπίσει τις ε, ε, διαδικασίες PAMS που είναι οι, τα φορητά συστήματα μετρήσεως εκπομπών που θα μας επιτρέψουν να επαληθεύσουμε τις εκπομπές. Το δεύτερο βήμα είναι να ορίσουμε ανώτατες τιμές, τιμές δηλαδή που δεν θα επιτρέπεται να υπερβαίνουν τα αυτοκίνητα, οχήματα. Και έτσι είναι το δεύτερο στάδιο αντιμετώπιση του προβλήματος. Τη δουλειά μας από εδώ και μπρος, πώς τη βλέπουμε. Από τις αρχές του 2016 θα θέλαμε να ξεκινήσουμε την παρακολούθηση και επαλήθευση οχημάτων και να ε, ε, ε, να εφαρμόσουμε το πρώτο σύνολο μέτρων που έχουν υιοθετήσει τα κράτη-μέλη από την αρχή του νέου έτους και να ορίσουμε τις ανώτατες τιμές, τις οριακές τιμές. Αυτό προτείνουμε σήμερα. Συζητούμε με τα κράτη-μέλη ποιες είναι αυτές οι τιμές που δεν επιτρέπεται να υπερβαίνουν οι εκπομπές και έχουμε επίσης και τα complementary boundary conditions, συμπληρωματικά οριακές συνθήκες, που έχουν να κάνουν με τον τρόπο της οδήγησης, με τις συνθήκες οδήγησης. Ε, ακολουθούν δύο συνεδριάσεις, Σεπτέμβριο-Οκτώβριο της Τεχνικής Επιτροπής, κατά τη διάρκεια των οποίων ελπίζουμε ότι θα είναι δυνατό να συζητηθούν και ενδεχομένω να εγκριθούν ή να συμφωνηθούν τα ανώτατα αυτά όρια. Το δεύτερο βήμα, όπως σας έλεγα που αποτελεί τμήμα της δέσμης 4 μέτρων που θα διαπιστώνεται και στο η πρώτη διαφάνεια. Το πρώτο στοιχείο για τις πραγματικές συνθήκε εκπομπών ε, προβλέπεται για το πρώτο τρίμηνο του 2016. Ιδιαίτερα όσον αφορά τις συγκεκριμένες τιμές σε περίπτωση των δοκιμών και Το 2016 προς το τέλος της χρονιάς αναμένεται να υιοθετηθεί το τελευταίο στατικό που έχει να κάνει με τις ε, δοκιμές συμμόρφωσης. Το τελευταίο στατικό των, ε, σε πραγματικές συνθήκες ε, εκπομπών οδήγηση. Και έτσι υιοθετείται μέχρι το τέλος του 2016 το σύνολο των μέτρων. Η υλοποίηση πώς μπορεί να προχωρήσει Τα όρια έχουν προσδιοριστεί από την νομοθεσία, αλλά δεν υπάρχει θέμα συζήτηση, αλλά σκεφτόμαστε ίσω την εισαγωγή ενδιάμεσων τιμών που θα επιτρέψει την προσαρμογή στο στάδιο που βρισκόμαστε των ε, οχημάτων και των κινητήρων που ήδη βρίσκονται στην αγορά και έτσι σιγά σιγά θα αποσυρθούν αυτά τα οχήματα και θα εισαχθούν τα απολύτως ε, κρίσιμα ανώτατα όρια, οι τιμέ δηλαδή που δεν μπορεί να υπερβαίνει ένα κινητήρα. Και όλα αυτά μέσα σε ένα κανονισμό. Αυτό που κοιτάμε βεβαίως αλήθεια είναι η υποχρέωση για πλήρωση των υποχρεώσεων του κανονισμού, αλλά και η ε, αντιμετώπιση βάρυνσης που θα σήμαινε η εισαγωγή των όρων αυτών για την αυτοκινητοβιομηχανία, να προσπαθούμε να εξορροπήσουμε και τους δύο, και τους δύο παράγοντες. Θεωρώ ότι μπορούμε να είμαστε αισιόδοξοι πως μέχρι το τέλος του έτους θα εξευρεθεί η συνένεση μεταξύ των κρατών μελών, με τα κρατημέλη προκειμένου να προσδοριστούν οι εκκρεμείς ακόμα παράμετροι. Αυτά ήταν όσα είχα να σας πω εισαγωγικά του θέματος και ευχαριστώ να ακούσω τις ερωτήσεις των βουλευτών. Σα ευχαριστώ λέει ο Πρόεδρος. Θα δώσω το λόγο στον επικεφαλής ε, της μονάδας ε, μεταφορών της ε, ΓΔΛΤΑ Κλίμα τώρα. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Καλημέρα σε όλους. Όπως και η Τζοάννα από την ΓΔΛΤΑ Γκρό θα σας ε, δείξω και εγώ κάποιες ε, διαφάνειες για να εξηγήσω το πλαίσιο, θυμίζοντας πού βρισκόμαστε σήμερα. Για το διοξίδιο του άνθρακα έχουμε την ε, διαδικασία ελέγχου NEDC, που είναι βέβαια από τη δεκαετία του 70, έχει, είναι κάποια ηλικία. Προσπαθούμε να εισαγάγουμε την WLTP, σχετικά με πιο αξιόπιστα και ακριβή δεδομένα εκπομπών διοξιδίου. Το 2014 συμφωνήσαμε σχετικά με, τις, με τα όρια και τις απαγορεύσεις και είχαμε συμφωνήσει ότι θα εισαχθεί το WLTP ως έλεγχος το συντομότερο δυνατόν. Σε συνεργασία λοιπόν με τους συνεργούς της Delta ε, Γκρό θέλουμε να εισαχθεί αυτή η δοκιμή μέχρι το Σεπτέμβριο του 2017 και για όλους τους τύπους οχημάτων μέχρι το Σεπτέμβριο του 2018. Ωστόσο, τα μέλη της Επιτροπής αυτής ε, που γνωρίζουν τις διατάξεις που αφορούν στα οχήματα, αυτό είναι το ένα σκέλος της προκλήσεως, διότι οι στόχοι διοξιδίου του άνθρακος για το 2015 και για το 2021 για τα ιδιωτικά αυτοκίνητα και τα βαν είναι, βασίζονται στις αξίες του NEDC. Ενώ εδώ βρισκόμαστε τώρα στον κύκλο εισαγωγής ε, του WLTP. Γιατί δοκιμάζοντας ένα όχημα με WLTP θα έχουμε υψηλότερες τιμές από αυτές που λαμβάνουμε μέσω του NEDC. Προσπαθούμε λοιπόν να καλύψουμε το θέμα αυτό μέσω της υφιστάμενης νομοθεσίας. Και με την υιοθέτηση και των δύο αναθεωρημένων κανονισμών υπάρχουν δύο τελογικές σκέψεις που δίνουν μια καθοδήγηση σχετικά με την συγκριτική αυστηρότητα, αν θέλετε να το ονομάσουμε έτσι, της, δηλαδή των οριακών τιμών για τους κατασκευαστές και για τους τύπους οχημάτων μετά την αλλαγή δηλαδή στη μεθοδολογία ελέγχου. Θα έπρεπε λοιπόν να έχουμε μια μελέτη συσχετισμού μεταξύ των κύκλων δοκιμής NEDC και WLTP. Και αυτά είναι αυτά επί των οποίων προσπαθήσαμε να δουλέψουμε τα τελευταία δύο χρόνια. Αυτή τη μελέτη δηλαδή συσχετισμού η οποία προσπάθεια Συσχετισμού είναι τεχνικώς εξαιρετικά περίπλοκη. Και επενδύσαμε πολλά όχι μόνο στο κοινό κέντρο ερεύνης και με τους συναδέλφους, αλλά είχαμε, πρέπει να πω, μεγάλη στήριξη και από τον κλάδο και από τα κράτη-μέλη, από τις αρμόδιες υπηρεσίες τις τεχνικές τους και από μη κυβερνητικούς οργανισμούς. Η μελέτη λοιπόν συσχετισμού τρέχει αυτή τη στιγμή θα εξακολουθήσουμε να εφαρμόζουμε τους στόχους NDC, αλλά οι μετρήσεις WLTP θα πρέπει να σχετιστούν στα μεγέθη που προκύπτουν από την NDC μέσω ενός εργαλείου που έχουμε αναπτύξει και το οποίο τελειοποιούμε αυτή τη στιγμή αλλά ελπίζουμε να είναι απολύτως λειτουργικό μέχρι το τέλος του έτους ώστε να μετατρέπουμε αν θέλετε τις τιμές NDC σε WLTP διατηρώντας όμως τις ε, ε, διατάξεις νομοθεσίας που αφορούν τα όρια NDC. Τώρα για την νομική υλοποίηση θα πρέπει να προχωρήσουμε προφανώς ε, εκ παραλίλου με τους συνέλφους της ΓΑΜΑΛΤΑΓΚΡΟ διότι είναι η νομοθεσία που θα πρέπει να εισαγάγει το, την, το τεστ WLTP υπό την έννοια των εκπομπών διοξιδίου του άνθρακος θα πρέπει ο κανονισμός να εξηγεί λεπτομερώς την ε, μεθοδολογία και αυτό θα πρέπει να το ψηφίσουν τα κράτη-μέλη στα πλαίσια της Επιτροπής Κλιματικής Αλλαγής και από εκεί και πέρα η Κομισιόν θα είναι εξοδοτημένη μέσω κατεξοδότηση πράξεως να το εφαρμόσει μέσω του παραρτήματος του κανονισμού. Και βεβαίως ε, ε, κατεξοδότηση πράξη με την επιφύλαξη όλων των ε, διατάξεων που τη διέπουν και με την έγκριση όλων των κρατών μελών. Όλα αυτά είναι μια περίπλοκη διαδικασία. Επαναλαμβάνω ότι ευχαριστώ όλους αυτούς που βοήθησαν στην προσπάθεια πάνω από όλα τους συναδέλφους της Γαμαλίτα ε, Γκρό και είμαι ε, στην απόλυτη διάθεσή σας για να απαντήσω ερωτήσεις σήμερα εδώ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Thank you very much. Ευχαριστώ πολύ. Να δώσουμε τώρα το λόγο στην Προεδρία του Συμβουλίου, ο κύριος Κριστόφ Χάνσεν, ε, περιβαλλοντικός ακόλουθος ε, της ε, μόνιμης αντιπροσωπείας του Λουξεμβούργου. Ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Πρόεδρε. Καλημέρα σε όλους. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω που μου δίνετε την ευκαιρία να σας ενημερώσω για τη διεξαγωγή των εργασιών στην ομάδα περιβάλλοντος στο Συμβούλιο για την μείωση των εκπομπών αερίων των οδικών οχημάτων. Δεν έχω την εντολή να μιλήσω εκ μέρους του Συμβουλίου. Μιλάω εκ μέρους μόνο τη της ε, Προεδρίας του Λουξεμβούργου. Στο πλαίσιο της ομάδας εργασίας ε, οι συζητήσεις οδήγησαν σε ένα συμβιβαστικό κείμενο υπό Ιταλική Προεδρία και επί Προεδρίας ε, συζητήσαμε στην ομάδα την έκθεση DES όπως επίσης και τις νομοδοτήσεις ΙΜΚΟ και ΤΡΑΝ. Οι αντιπροσωπείες έλαβαν γνώση των απόψεων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σε σχέση με ε, τους ε, δείκτες αλλαγής ταχυτήτων και τους μετρητές κατανάλωσης καυσίμου και το Συμβούλιο όπως και το Κοινοβούλιο έχουν κάποια, κάποιες, κάποιους ενδιασμούς σε σχέση με τις κατεξοδότηση πράξης για τον, ορισμό, ε, για τον καθορισμό των οριακών τιμών γιατί το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα ήθελε μάλλον μια τακτική νομοθετική διαδικασία. Ε, επίσης θα θέλαμε να υπάρξουν ε, διευκρινήσεις από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τον ενδεχόμενο αντίκτυπο της RDE ε, για την πρόταση κανονισμού και επίσης για τις εξελίξει στο πλαίσιο της Τεχνικής Επιτροπής ε, για τα μηχανοκίνητα οχήματα, τις οποίες προεδρεύει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ε, προβλέπεται για την επόμενη εβδομάδα η συνεδρίασή της και μόνο μετά τη συνεδρίαση αυτή θα μπορέσω να σας δώσω περισσότερες πληροφορίες. Εν τω μεταξύ μπορώ να σας διαβεβαιώσω ότι η Προεδρία του Λουξεμβούργου αναμένει εναγωνίως ε, τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας 23 23η Σεπτεμβρίου της Επιτροπής Περιβάλλοντος για την έκθεση για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε στις διαπραγματεύσεις μας με το Κοινοβούλιο ευχαριστώ πολύ. Με ευχαριστώ πάρα πολύ. Αρχίζω τον κατάλογο των ομιλητών με τον Καρλ Χάινς Φλόρενς. Καταρχάς, θα ήθελα να ευχαριστώ τους δύο εκπροσώπους της Επιτροπής. Παρακολουθώ και εγώ εδώ και μερικά χρόνια. Το θέμα αυτό είναι αμφίβολα, πάρα πολύ δύσκολο. Υπήρχαν μια σειρά από βρώμικα κόλπα, εσκεμμένες δηλαδή κινήσεις των πρωταγωνιστών προκειμένου να ε, αλλοιωθούν οι τιμές. Εκτιμώ ιδιαίτερα τοποθετήσει του εκπρόσωπου του Λουξεμβούργου. Αντιλαμβάνομαι ότι εκπροσωπεί το Λουξεμβούργο, αλλά αυτό που έχω να πω τους έχω εδώ στο Κοινοβούλιο, δουλειά σας δεν εκπροσωπείστε το Μεγάλο Δουκάτο, αλλά το Συμβούλιο, στο οποίο εδρεύουν και συνεδριάζουν μεγάλα αυτοκίνητο παραγωγά κράτη. 8.000 αυτοκίνητα παράγονται κάθε χρόνο, κυκλοφορούν στους δρόμους της Ευρώπης κάθε χρόνο. Άρα δεν μπορούμε να έχουμε πιο ευέλικτες τιμές, αλλά πιο αυστηρές τιμές. Και αυτό όχι γιατί θέλει, δεν θέλουμε να αποδειχθεί ότι πως έχουμε δίκιο ή να επικρατήσει το δικό μας, αλλά γιατί πρόκειται για την υγεία των πολιτών. Και να πω και κάτι για, τα, ε, για το κόστος. Θυμάστε τι είδους ε, αντιδράσεις και τι τσίρκο είχε προκύψει όταν μιλούσαμε για κατώτατε τιμές. Ήταν μια απόλυτη ανοησία κάθε δυνατότητα εξοικονόμησης από τα νεοπαραγόμενα αυτοκίνητα σε δύο-τρία κράτη οδήγησαν σε εκρηκτική αύξηση των τιμών με την εισαγωγή νέων καυσίμων. Γι' αυτό λοιπόν θα λέω στην Επιτροπή ότι πρέπει πια να σταματήσει αυτή η ιστορία. Είναι πια χιλιάδες οι πρόσωποι των λόγων που κυκλοφορούν μέσα στα κτίρια. Α σταματήσει λοιπόν αυτή η ιστορία. Δεν θέλουμε να καταστρέψουμε την αυτοκίνητο βιομηχανία μας, κατηγορείται για κάτι τέτοιο, αλλά δεν είναι ε, δεν υπάρχει καν κίνδυνο να καταστραφεί αυτό το αυτοκινητοβιομηχανία γιατί είναι στο ισχυρότερο σημείο τη αυτή τη στιγμή στην ανάπτυξη της στην Ευρώπη. Α γίνει λοιπόν αυτό που ζητεί το Κοινοβούλιο προκειμένου να έχουμε σωστέ οριακέ τιμέ. Και θα έλεγα κύριε εκπρόσωπε του Συμβουλίου ότι αντιλαμβανόμαστε πώ δεν θέλουν τα κράτη τη καταξιοδότηση πράξη, αλλά έχουμε καταφέρει χάρη στις καταξιδότητες πράξεις να ε, αναγκάσουμε την Επιτροπή και το Συμβούλιο να ανακρούσουν πρίμνα και να κάνουν επιλογές διαφορετικές από τις αρχικές τους. Γι' αυτό λοιπόν και πρέπει να κάνουμε κινήσεις για να στηρίξουμε και την αυτοκίνητο βιομηχανία, γιατί και μέρα μου αρέσουν να μπαίνω σε αυτοκίνητο και να κάνω βόλτες. Ευχαριστώ κύριος Χρότε. Ναι. Και εγώ θα μπω σε ένα θέμα που έχει να κάνει με εξοικονόμηση χαρτιού κυρίως, γιατί στις οριακές τιμές έχουμε δει άνευ προηγουμένου ψέματα και παραπλάνηση. Πραγματικά είναι πολύ δυσάρεστη κατάσταση με την εισαγωγή των ορίων του διοξιδίου του άνθρακα ευρωπαϊκά όρια 5 και 6, Euro 5 και Euro 6. Ε, ακούστηκαν διάφορα φοβερά πράγματα και τάχα ότι θα παρακολουθούσαμε με άγρυπνο μάτι τις ε, δοκιμές. Εδώ όμως βλέπουμε ότι και οι κοινοτικές αρχές, οι δημοτικές αρχές δίνουν τη δυνατότητα να επαληθεύσουν ε, τι συμβαίνει. Βρίσκονται υποπίεση όσον αφορά την διαφύλαξη των, ε, της ποιότητας του ατμοσφαιρικού αέρα και πρέπει να τους επιτραπεί να επαληθεύουν σε πραγματικούς όρους και όχι με συνθήκες εργαστηρίου, με τους καλύτερους δυνατούς ε, μηχανολόγους και με τις καλύτερες δυνατές συνθήκες που άλλωστε ξέρουμε ότι μπορούν να ε, παραβιάσουν ή να παραχαράξουν τα αποτελέσματα των δοκιμών ε, η αυτοκινητοβιομηχανίας γιατί πρέπει να γνωρίζει ο πολίτης με τι είδους ρήπους επιβαρύνεται. Αυτά τα κόλπα πρέπει να σταματήσουν με κάθε και με διάφορα άλλα πράγματα μπορούν να χρησιμοποιούν και σχέση με τις ε, εξουσιοδότηση πράξεις θα κοιτάμε και την τελευταία τελεία και κόμμα δεν πρόκειται να επιτρέψουμε να παραβιαστούν οι όροι. Εφόσον δεν πληρούνται οι προποθέσεις που έχει δώσει το Κοινοβούλιο δεν θα προχωρούν. Και έχουμε δει ε, αδιεξόδους στους τριμερείς διαλόγους, τα ξέρετε κι εσείς αυτά. Έχουμε δει συνεδριάσεις τριμερούς διαλόγου που έχουν κρατήσει μόλις 30 δευτερόλεπτα γιατί δεν υπήρχε κανένα πεδίο συζήτησης. Επίσης, πρέπει να κοιτάξουμε τα ηλεκτρικά οχήματα. Εάν ε, δηλαδή μπορούμε να προωθήσουμε σαν λύση πιο ε, οικολογική τα ηλεκτρικά οχήματα και αν είναι το ίδιο το να χρησιμοποιούμε ένα οικολογικό όχημα στην ε, Σουηδία, τη Γερμανία που 25% ηλεκτρικό από την αιωλική ενέργεια ή την Πολωνία και πόσο μπορεί να επιβαρύνει το περιβάλλον η χρήση τους ανάλογα με την προέλευση του ηλεκτρικού. Όλα αυτά λοιπόν και επανέρχομαι για να πω ότι πρέπει να παρακολουθείτε με κάθε ακρίβεια ο κύκλος της δοκιμής χωρίς παραβιάσεις που φτάνουν στο 25-30% από ό,τι βλέπουμε τώρα. Για τα 130 γραμμάρια εκπομπών που μας αναφέρεται για το διοξείδιο του άνθρακα έχουν να κάνουν μια εξαιρετικά οικονομική οδήγηση η οποία δεν αντιστοιχεί σε καμία πραγματικότητα στους ευρωπαϊκούς δρόμους. Παρακαλώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ και ευχαριστώ για τις παρουσιάσεις. Εμένα το ενδιαφέρον μου είναι γενικό αλλά και πολύ συγκεκριμένο ε, επειδή είμαι εισηγήτρια για την οδηγία NEDC ε, και ήταν εξ αρχής ένα πάρα πολύ σημαντικό ζήτημα. Θυμάμαι την αρχική ανεπίσημη παρουσίαση που άκουσα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, για το, από το τμήμα ποιότητας του ατμοσφαιρικού ε, αέρα. Υπήρχαν κάποια θέματα συμβατότητας ε, για το Euro 4, ε, μετά μιλούσαμε για το Euro 5 και τώρα μιλάμε για το Euro 6 και σε κάθε μία από αυτές τις συζητήσεις και πριν από το Euro 4 ήταν σαφές ότι υπήρχε τεράστιο χάσμα μεταξύ της πραγματικής απόδοσης και της απόδοσης ε, που ε, αποτελεσματικά κατέγραφαν οι διαδικασίες δοκιμών που ε, ίσχυαν και εξακολουθούν να ισχύουν. Ένα πράγμα το οποίο με μπερδεύει είναι πώς είναι δυνατόν ε, για μεγάλο τμήμα ε, δεκαετιών να συνεχίζουμε με αυτή τη διαδικασία παρόλο που ξέρουμε ότι η ρήπη είναι διαφορετική από αυτούς που καταγράφονται ε, δεν έχει σημασία τώρα να αρχίσουμε να κατηγορούμε ένα τον άλλον γιατί αυτό δεν θα μας οδηγήσει πουθενά αλλά καταλαβαίνω ότι ε, επικεντρωθήκαμε περισσότερο στον άνθρακα και λιγότερο στον τομέα των ρήπων. Τώρα λοιπόν αυτή τη στιγμή έχουμε φτάσει μια κατάσταση, πρέπει να το αντιμετωπίσουμε αυτό το πρόβλημα, γιατί ένα μεγάλο μέρος των ζητημάτων που έχουμε να καλύψουμε ε, όταν εξετάζουμε την οδηγία είναι ότι υπάρχουν δήμοι στην Ευρωπαϊκή Ένωση που είναι έτοιμοι, ε, τουλάχιστον το Λονδίνο, υπάρχουν τόσα πολλά φιλόδοξα σχέδια για να εξασφαλιστεί ότι θα βελτιωθεί η δημόσια ισχύ και δεν μπορούν να τα πραγματοποιήσουν γιατί δεν ε, ε, είναι σίγουροι ότι, ε, ότι μπορούν να αποφασίσουν ποιο όχημα μπορεί να επιτρέπεται σε κάποια ζώνη, γιατί δεν μπορούν να αποφασίσουν, ε, δεν, δεν μπορούν να αποφασίσουν βάσει της, της συμβατότητας Euro 5 και Euro 6, δεν ξέρουν ακριβώς τι πρέπει να κάνουν. Όλοι το γνωρίζουμε όμως αυτό, ε, έχουμε γνώση του προβλήματος αυτού, ε, πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα υπάρχει το πρόβλημα, αλλά πώς θα προχωρήσουμε. Και το δικό μου ενδιαφέρον επικεντρώνεται στο εξή. Ή πρέπει στην οδηγία να μην συμπεριλάβουμε ανώτατα όρια τα οποία δεν είναι ε, υπερ, υπερβολικά φιλόδοξα, αλλά όχι και πολύ λίγο φιλόδοξα. Ε, πρέπει να ε, συνεισφέρουμε και για να το κάνουμε αυτό πρέπει να ξέρουμε τα χρονοδιαγράμματα. Μιλάμε για το 2019 το 2019 θα έχουμε πλήρη συμβατότητα, αν δούμε τους συντελεστές συμβατότητας που προτείνονται και θα έλεγα ότι αυτό δεν είναι αρκετό. Νομίζω λοιπόν ότι το μήνυμα που πρέπει να στείλουμε με τη συζήτηση αυτή, μόνο μια συζήτηση είναι, να ζητούσουμε λοιπόν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τα επίπεδα συμβατότητας ε, να απορρίψουν τα υψηλά ε, επίπεδα συμβατότητας που ζητά η βιομηχανία. Ε, το ξέρουν εδώ και πάρα πολύ καιρό. Μπορούν να το κάνουν, εκείνοι λένε ότι δεν μπορούν. Απλώς πρέπει να ενθαρρυνθούν να το κάνουν πιο γρήγορα. Λοιπόν, να μην πούμε λοιπόν ε, ε, συντελεστή συμβατότητας 1,5 ε, για παράδειγμα, ε, ξέρω ότι υπάρχουν προβλήματα, αλλά ίσως θα έπρεπε να πιέσουμε λίγο περισσότερο στις συνομιλίες μας με τη βιομηχανία. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Κύριος Γέρπαρτ. Ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα να ευχαριστήσω την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τα εναρκτήρια σχόλιά της. Ε, θα ξεκινήσω με ένα γεγονός. Το γεγονός είναι ότι μας κορόιδεψαν ε, και τα 500 εκατομμύρια ε, πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης παραπλανήθηκαν επίσης για τα αποτελέσματα των δοκιμών αυτών των οχημάτων και αν σε κοροϊδεύουν για τόσο μεγάλο χρονικό διάστημα θα έπρεπε να είναι υποχρέωσή μας να το αποκαταστήσουμε το πρόβλημα το συντομότερο δυνατόν και να επανέλθουμε σε ε, δοκιμές ε, για την παραγωγή εκπομπών σε πραγματικές συνθήκες οδήγησης. Βλέποντας το χρονοδιάγραμμα ε, σκέφτομαι ότι δεν χρειάζεται να κάνουμε πλέον τίποτε γιατί τα έχουμε όλα έτοιμα αυτή τη στιγμή. Έχουμε ηλεκτρικά ε, οχήματα που έχουν επεκταθεί και καλύπτουν μεγάλο τμήμα του στόλου μας. Παρ' όλα αυτά χρειαζόμαστε κάποιο επίπεδο φιλοδοξία. Δεν θα επαναλάβω αυτά που είπαν οι συνάδελφοι γιατί συμφωνώ απολύτως μαζί τους. Δύο πολύ συγκεκριμένες ερωτήσεις έχω να απευθύνω στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Πρώτη ερώτηση. Για ποιο λόγο Γενική ε, Διεύθυνση Ανάπτυξης ε, είναι υπεύθυνη για το θέμα αυτό, βλέποντας ε, ε την ε, το, ιστοσελίδα της, ε, ε οι πρώτες φράσεις είναι «εργαζόμαστε για την ανάπτυξη». Μα εδώ όμως δεν μιλάμε για αυτό το θέμα, μιλάμε για την ύπαρξη πραγματικών συνθήκων, για για την καταγραφή των εκπομπών σε πραγματικές συνθήκες οδήγησης και τέτοιου είδους διαδικασίες δοκιμών. Ε, η, η Επιτροπή ΕΜΒΗ είναι υπεύθυνη για το θέμα αυτό ε, στο Κοινοβούλιο, το οποίο μου φαίνεται λογικό. Ίσως θα μπορούσε να μας εξηγήσει λοιπόν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή γιατί τέτοιου είδους κατανομή εργασία στο πλαίσιο της Επιτροπής. Κάτι ακόμη για τα αυτοκίνητα που κινούνται με ντίζελ, όπως επίσης και τα οξύδια του αζότου. Ε, σύμφωνα με ε, μελέτες του κοινού ε, κέντρου ερεύνης και άλλων φορέων υπάρχει παραβίαση από, από, τα, από τα 6 στα 9 αυτοκίνητα των επιπέδων, των οριστέντων επιπέδων. Πώς πρέπει να τα μειώσουμε, έχετε σκοπό να μειώσετε τις παραβιάσεις αυτές ε, στο μηδέν, γιατί αυτό είναι που θέλουμε να επιτύχουμε με τη νέα αυτή διαδικασία δοκιμών, η παραβίαση να πάει σε μηδενικό επίπεδο και να σταματήσει ε, το συντομότερο δυνατόν αυτή η λάθος ε, δοκιμασία, διαδικασία δοκιμών. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ Πρόεδρε, ευχαριστώ την Κομισιόν και τους εκπροσώπους τη που μας εξήγησαν πού βρισκόμαστε στη διαδικασία τι μπορούμε ακόμα να περιμένουμε και τι μπορούμε να συζητήσουμε, αλλά είναι σαφές από αυτές τις παρεμβάσεις ε, τουλάχιστον ότι για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι πολύ σημαντική αυτή η διαδικασία, παρακολουθούμε στενά και προσεκτικά και ακούγοντας ε, τους συναδέλφους είναι ικανοποιητικό να ακούμε τα στοιχεία αυτά γιατί ίσως και κάποια χώρα και ίσως και σημαντική χώρα Ματίας να διαδραματίζει πολύ σημαντικό ρόλο στη διαμόρφωση των στοιχείων αυτών. Είμαστε έτοιμοι να απορρίψουμε ένα αποτέλεσμα των διαπραγματεύσεων που θα θεωρήσουμε αρνητικό. Γιατί έτσι φαίνεται να πηγαίνει. Επίσης, είναι απογοητευτικό να βλέπουμε ότι ο αυτοκινηστικός κλάδος ξανά και ξανά προσπαθεί να κατεβάσει τα όρια. Γνωρίζουμε τη μάχη που εδόθη για να πάμε στην παρούσα νομοθεσία και γνωρίζουμε πόσα χρόνια λειτουργούν άσχημα και ελλειπώς οι δοκιμές αυτές. Τώρα κάνουμε κάτι για τις δοκιμές και βεβαίως ο κλάδος ζητάει χρόνο προσαρμογής γιατί δυσκολεύεται. Με συγχωρείτε αλλά εδώ πέρα δεν έχουν επικαιροποιηθεί όλα αυτά, όλες αυτές οι δοκιμές εδώ και πάρα πάρα πολλά χρόνια. Πρέπει να είμαστε πολύ πιο αυστηροί στον χρόνο που θα τους δώσουμε. Για να φτάσουμε, εν πάση περιπτώσει, σε μια συμμόρφωση. Τώρα για, το, για τα οξύδια του αζότου. Μια ερώτηση προς την Κομισιόν. Γνωρίζω ότι τώρα συζητούμε αυτά τα, αυτούς τους παράγοντες, τους συντελεστές σχετικά με τη συμμόρφωση. Πώς μπορούμε διαφορετικά να τους δούμε παρά μόνον ως μικρότερους στόχους από αυτούς που είχαμε θέσει. Είχαμε θέσει ένα σαφέστατο στόχο 80 το Σεπτέμβριο του 2014. Αν όμως δουλεύουμε επί στόχων και το συζητούμε, σημαίνει ότι επιτρέπουμε υψηλότερες ε, εκπομπές ρήπων. Δηλαδή δεν συμμορφωνόμαστε προς την υφιστάμενη νομοθεσία. Και αυτό σημαίνει ότι παρακάμπτουμε την νομοθεσία κατά την άποψή μου. Εφόσον συζητούμε για conformity factors, σημαίνει ότι αυτός ο συντελεστής θα πρέπει να πάει στο 1, για να πάμε δηλαδή στα επίπεδα που είχαμε συμφωνήσει ως συνομοθέτες. Και με αυτό το συντομότερο δυνατό. Επομένως ερώτηση προς την Κομισιόν, τι συντελεστές επεξεργάζεστε και πότε θα σταματήσουν αυτοί οι συντελεστές να ισχύουν. και γνωρίζω ότι ο κλάδος αυτοκινηστικός συζητάει 2,75 συντελεστή, δηλαδή περί τις τρεις φορές τα όρια που είχαμε συμφωνήσει και αυτό να παραταθεί για πολλά χρόνια επίσης. Άρα λοιπόν, εγώ θα ήθελα να ακούσω από την Κομισιόν ότι αυτοί οι συντελεστές θα εφαρμοστούν για πολύ πολύ σύντομο χρονικό διάστημα, για να πάμε σε συντελεστή 1 σε maximum 4 χρόνια, και ότι δεν θα είναι αυτοί οι συντελεστές υψηλότεροι του 1,5 για το διάστημα προσαρμογής. Αυτό θα ήθελα να ακούσω από την Κομισιόν και ότι θα εφαρμοστεί το συντομότερο δυνατό. Άλλη ερώτηση. Μας είπατε ότι αυτή τη στιγμή υπερβαίνουμε τα, τα όρια των ε, οξυδίων του αζότου και υπάρχουν διάφορες χώρες που επιτρέπουν υψηλότερους συντελεστές συμμόρφωσης που σημαίνει ότι έχουμε μεγαλύτερη υπέρβαση των εκπομπών ε, οξυδίων του αζότου. Για 10 χώρες. Πόσες περισσότερες χώρες θα υπάρχουν στον κατάλογό σας όσο υψηλότερου συντελεστέ αποδέχεστε. Υπάρχει άμεση διασύνδεση και είμαι βέβαιος ότι τη γνωρίζετε και πώς λειτουργεί. Θα ήθελα λοιπόν να ακούσω από την Κομισιόν πότε ο συντελεστής αυτός θα φτάσει στο 1 στη μονάδα. Αυτά για τα ντίζελ και τα οξύδια του αζότου. Τώρα για το διοξείδιο του, άνθρω του άνθρακα. Συγκρίσιμη αυστηρότητα, μάλιστα. Αν πάμε από παλαιά δοκιμή σε νέα δοκιμή χρειάζεται μελέτη σχετισμού κτλ. Μέχρι εκεί σας παρακολουθώ. Αλλά τότε η ερώτησή μου είναι ποιους συντελεστές συμπεριλαμβάνεται σε αυτή τη μελέτη σχετισμού. Ποιος είναι δίκαιος συντελεστής μεταξύ της παλαιάς μεθόδου και της νέας μεθόδου ώστε να συμπεριλάβουμε αυτήν την μετάβαση ποια είναι δηλαδή μια δίκαια ευελιξία που πρέπει να εφαρμοστεί και σε ποια σημεία απλώς αντιγράφεται ανόητα, ανόητες διατάξεις της προηγούμενης δοκιμής. Γιατί τώρα δουλεύετε επί τη βάση νέας δοκιμής αλλά μέσω της ε, μελέτης σχετισμού επαναλαμβάνεται τις ίδιες ανοησίες που είχαμε παλαιότερα και τώρα. Εγώ δεν θέλω μέσα την εξωτερική φόρτιση της μπαταρίας, δεν θέλω αυτούς τους παράγοντες και τους συντελεστές που βλέπω στην ε, σχετισμό. Γιατί αυτά ε, περιείχε η παλαιότερη μέθοδος δοκιμής. Γιατί τα συμπεριλαμβάνεται στη νέα μέθοδο. Θα ήθελα να ακούσω από εσά ότι αποκλείεται τους παράγοντες αυτούς και ότι πάτε στην ταχύτερη δυνατή υλοποίηση. Και το πιο σημαντικό από όλα, από το 2025 όταν θα έχουμε νέα πρότυπα για τις εκπομπές των οχημάτων, θα σταματήσουμε με αυτή τη μελέτη σχετισμού. Δηλαδή συγκρίσιμη αυστηρότητα, διότι ιδάλλως αυτό θα σημαίνει στην πραγματικότητα ότι είμαστε το ίδιο ελαστικοί όσο ήμασταν πάντοτε. Θα πρέπει μόνο επί τη βάση της νέας μεθόδου δοκιμής να εφαρμόζουμε τα όρια. Και τελευταία ερώτηση. Θα λάβετε με κάποιον τρόπο υπόψη σας αυτά τα super credits. Δηλαδή, εκεί που εφαρμόζεται η παλιά μέθοδος. Δηλαδή, σε ποιο τύπο οχήματος δίδεται super credits σε ποιες από αυτές τις περιπτώσεις θα εφαρμόζεται η παλαιά μέθοδος και από ε, αυτού θα ήθελα μια σαφή απάντηση από εσά. Ιδάλλως το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα αναλάβει μια πολύ αυστηρή προσέγγιση. Σας ευχαριστώ κυρία Τζορντάνο. Ντονάνο. Euh, σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ και την ε, Κομισιόν για τις εξηγήσεις που μας έδωσε. Σύμφωνα με τη νέα μέθοδο θα έχουμε ακριβέστερα όρια υποτίθεται και θα έχουμε και μια διαφάνεια την οποία δεν μπορώ παρά να χαιρετήσω. Αλλά θα ήθελα να επικεντρωθώ στο εξή. Η προσαρμογή του αυτοκινητικού κλάδου και των, αυτοκιν... και των παραγωγών ενέχει και άλλους τομείς. Υπάρχουν και ενώσεις καταναλωτών που ανησυχούν για την επεξεργασία αυτή που κάνετε για τις μεθόδους δοκιμής. Και έχω δύο ερωτήσεις. Η Κομισιόν έχει επικαιροποιημένη πρόσφατη μελέτη σχετικά με το σεβασμό των ορίων για το 2020 για τον ε, κλάδο τον, τον αυτοκινηστικό. Και δεύτερον, από το input που είχατε από τους Αμερικανούς κατασκευαστές ε, και ειδικού στα πλαίσια της TTIP και των ελεύθερων συναλλαγών, ποια είναι η, ποιο είναι το συγκριτικό πλεονέκτημα των Ευρωπαίων κατασκευαστών και πώς θα μπορούσαμε να το διατηρήσουμε αυτό μακροπρόθεσμα. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ κυρία Σίβη. Ευχαριστώ πρόεδρε. Εγώ συμφωνώ απόλυτα με αυτά που είπε ο συνάδελφος των Πρασίνων και με τις απορίες γενικώ που εξέφρασαν οι συνάδελφοι. Και αυτό που θα ήθελα να θυμίσω και δεν πρέπει να το ξεχνούμε ποτέ αφορά τον όγκο των εκπομπών που υπολογίζουμε στο 3% για τις αστικές περιοχές και οι δεκάδες χιλιάδων πρώιμοι που οφείλονται στη ρήπανση και στη μόλυνση και το σχετικό κόστος για την υγεία από όλους αυτούς τους πρώιμους θανάτους Δηλαδή αυτή είναι μια σωστή βάση και σωστό πλαίσιο για να συζητήσουμε για τις προϋποθέσεις και για τα επόμενα βήματα που θα πρέπει να αναλάβουμε προς τις διατάξεις αυτές. Είναι θεμελιώδους σημασία το ότι εδώ συμφωνούμε σε θεωρητικό επίπεδο για την προστασία της δημόσιας υγείας να ακολουθείτε από εξακρίβωση, από έλεγχο και ο ρόλος των ελεγκτών θα πρέπει να αναλαμβάνεται και από την ε, Κομισιόν ώστε να μην παράγονται κενά και παραθυράκια στην υλοποίηση της νομοθεσίας. Και έχουμε και ένα στρεβλωτικό χαρακτήρα αυτή της έννοια της ευελιξίας που παραχωρείται και που αναφέρθηκε και παραχωρείται στον αυτοκινητικό κλάδο σχετικά με τους ατμοσφαιρικούς ρήπους που έχει επιφέρει στρέβλωση και στην ουσία ελάττωση των στόχων που είχαμε θέσει για τις τιμές αναφορές. Και χωρίς να επαναλάβω τα όσα είχαμε ήδη πει για τους νέους μηχανισμούς ελέγχου και για το διοξείδιο του άνθρακος και για τους υπόλοιπους ρήπους, εμένα με ανεσοχούν ιδιαίτερα οι πιέσει που ασκούνται από τους κατασκευαστές, από τον κλάδο, σε αυτήν την εισαγωγή των στοιχείων ευελιξίας. Γιατί δεν μπορεί να δεχθεί κανείς ότι στην ευθυγράμμιση των στόχων προς τα νέα κριτήρια, στην ουσία θα ελαττώσουμε θα αποδυναμώσουμε τα όρια μεγίστων εκπομπών που είχαμε θέσει νωρίτερα. Πρέπει επίσης να υπογραμμίσουμε ότι για μία ακόμα φορά βρισκόμαστε σε μία διαδικασία κατά την οποία οι συνομοθέτες βρίσκονται σε απόλυτη αδυναμία ή μάλλον να το πω έτσι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή στα πλαίσια της Επιτροπολογίας αποκλείεται από την ενεργό συμμετοχή που πρέπει να έχει σε αυτή την αναθεώρηση. Θα πρέπει οπωσδήποτε να διαδραματίζουμε έναν πολύ πιο ενεργή ρόλο από αυτόν που μας έχει παραχωρηθεί στην πραγματικότητα. Θα ήθελα λοιπόν να ζητήσω από την Κομισιόν να εξασφαλίσει η προσαρμογή των μεθόδων θα γίνει κατά τρόπον ώστε οι, τα 95 χιλιόγραμμα να τηρηθούν για το 2025 χωρίς κανενός είδους ευελιξία και ότι από το 2017 ε, για τα οξύδια του αζότου δεν θα έχουμε μεγαλύτερο συντελεστή από 1,5 σχετικά με την ευελιξία αυτή και τελικά θα πρέπει να μειωθεί στο 1 όπως ήδη είπε ο συνάδελφος από το 2019. Και από το 2020 θα πρέπει όλα αυτά να εφαρμοστούν για όλους τους τομείς οχημάτων που ορίστηκαν όρια. Σας ευχαριστώ και εγώ, λέει ο πρόεδρος, ο κύριος Ιβο Μπένετ. Πρόεδρε, ευχαριστώ και θα είμαι σύντομο. Ύστερα από όλες αυτές τις εισαγωγές, ευχαριστώ την Επιτροπή και το Σύμβουλο, την Προεδρία για τα όσα μας είπαν εισαγωγικά. Θα ήθελα κάποιες συγκεκριμένε ερωτήσεις να διατυπώσω. Καταρχάς, όσον αφορά την απόκληση μεταξύ των πραγματικών επιδόσεων και εκείνων που καταγράφονται στις δοκιμές από τα έγγραφα. Κυρίως ε, αυτά που βλέπουμε από τις μεταφορές και το περιβάλλον. Έχουμε αύξηση αυτής της απόκλησης στο 40%. Μπορεί η Επιτροπή να μας επιβεβαιώσει αυτό το νούμερο. Επίσης, για το WLTP και τις ευελιξίες που αναφέρθηκαν και νωρίτερα, και φαντάζομαι ότι και εμείς πάλι από το Transport and Environment ε, έχουμε τις ίδιες πηγές με τον συνάδελφο. Πολύτιμη πηγή. Μπορεί η Επιτροπή λοιπόν να μας επιβεβαιώσει ότι υπάρχει τέτοια ευελιξία. Που ασφαλώς επηρεάζει και θα επηρεάσει. Θα μπορούσε άλλωστε και να υποβαθμίσει σημαντικά την τήρηση των στόχων που είναι νομοθετική. οξίδια του αζότου και διοξίδιο του αζότου, που ξέρουμε ότι είναι οι πιο επιβαρυντικοί παράγοντες και προξενούν και προώρους θανάτους λόγω της κακής ποιότητας του ατμοσφαιρικού αέρα. Εντάξει, μπορούμε να καταλάβουμε ότι μπορεί να υπάρχει μια σταδιακή εισαγωγή των ε, τιμών, η δυνατότητα προσαρμογής δηλαδή. Αλλά όπως ρώτησε και η συνάδελφος νωρίτερα, τι είδους λογική προσαρμογής θα προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή περίοδο 1 ως 1,5 έτους, συντομότερη, μεγαλύτερη και πώς θα εξασφαλίσει ότι δεν θα ε, υποβαθμιστεί η τήρηση αυτών των στόχων. Άλλωστε θα πρέπει πρόεδρε για να καταλήξω ότι αυτές οι δοκιμές σε πραγματικές συνθήκες των εκπομπών να συμπεριλαμβάνουν και θέλω να το επιβάσω αυτό η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τις εκπομπές μικροσωματιδίων. Γιατί και αυτό είναι εξίσου σημαντικό με το άζωτο, με τα οξύδια του άζωτου. Um, Κυρία Νταγή, ευχαριστώ. Ευχαριστώ την Επιτροπή, ευχαριστώ το Συμβούλιο για τις εγωγικές του τοποθετήσεις. Θέλω κι εγώ μαζί με τους συναδέλφους να υπογραμμίσω τη σημασία που αποδίδει το, το Κοινοβούλιο και η Επιτροπή μας στην αυστηρή τηρήση των όρων ε, των νομοθετημάτων που ισχύουν ήδη. Σε αυτό επιμένουμε ιδιαίτερα. Το μήνυμα πρέπει να περάσει τόσο στην Επιτροπή όσο και στο Συμβούλιο γιατί σε τελευταία ανάλυση εδώ μιλάμε για την επιβάρυνση της υγείας των πολιτών μας. Και αν συμβιβαστούμε σε χαμηλότερο επίπεδο προστασίας, επιβαρύνουμε, θέτουμε σε κίνδυνο την υγεία και τη ζωή των πολιτών μας. Ερωτήσει λοιπόν κυρίως προς την Επιτροπή. Εθίγημένα, αλλά θα ήθελα ιδιαίτερα να υπογραμμίσω γιατί θα ήθελα απάντηση να δοθεί ξεκάθαρη στο ζήτημα το οποίο άλλωστε θα κρίνει και το πλαίσιο μέσα στο οποίο θα κινηθούν οι προτάσεις. Εάν λοιπόν η Επιτροπή εισάγει παράγοντες συμμόρφωσης, όπως λέγεται. Μπορεί πιο συγκεκριμένα να υποδείξει τι είδου παράγοντες συμμόρφωσης σκοπεύει να επιλέξει και σε ποια στάδια ή με πόσα στάδια σκοπεύει να τους εισαγάγει. Γιατί κάθε φορά που εισάγεται παράγον ε, προσαρμογής, ξέρουμε ότι υποβαθμίζεται η τήρηση των νομοθετικά ορισμένων όρων. Και όταν γίνει αυτό, πώς μπορεί η Επιτροπή να εξισορροπήσει με μέτρα το γεγονός ότι αστικά κέντρα και κόμβοι μπορεί να έχουν και διπλασιασμό ακόμη των υπερβάσεων των ανώτητων ορίων. Επίσης ε, επιμένω στο ότι σήμερα υπάρχει ένας ε, στόχος, καλός στόχος μεν, αλλά ανεπαρκές σύστημα δοκιμών της στήριξης του. Πώς η Επιτροπή με τα νέα μέτρα θα αποφύγει κατάσταση κατά την οποία θα μπορούσαμε να έχουμε αποτελεσματικές δοκιμές σε πραγματικές συνθήκες, αλλά αποδυναμωμένους όρους και οριακές τιμές. Τελική ερώτηση. Η Επιτροπή έχει στόχο την τροποποίηση του, των δοκιμών όπως προτείνονται τώρα σε πραγματικές συνθήκες εκπομπών για τα οξύδια του αζότου έτσι ώστε να συμπεριλάβουν και άλλες εκπομπές. Ευχαριστώ για άλλα σέντερ. Ευχαριστώ πρόεδρε. Ε, και εγώ θα συμφωνήσω με τον συνάδελφο τον Ματίας Γκρότε και θα ήθελα να μας εξηγήσει η Κομισιόν. Μας είπε ο εκπρόσωπος της Ένβι ε, ότι εμπάσχετος βρίσκονται στη συνεργασία με την ε, ΓΔ Ανάπτυξη, αλλά θα ήταν πολύ σημαντικό μετά από όλα αυτά που αναλύσαμε, είδαμε, ακούσαμε σχετικά με τις ε, παραβιάσεις σχετικά με τις εκπομπές, γιατί έχουμε, τα έχουμε δει αυτά τα πράγματα η πραγματικότητα δεν ανταποκρίνεται σε αυτά που γράφουμε στο χαρτί, τα θεωρητικά. Δηλαδή, ρωτώ την Κομισιόν, πώς τελικά θα μπορέσουμε να επιβάλλουμε ένα πλαίσιο κανονισμών που να έχει μία συνένεση, διότι ο κανένας μπορεί να έχει τις επιθυμίες του και τα όνειρά του, αλλά αν έχουμε πόλεμο με τη βιομηχανία, γιατί αυτό συμβαίνει κάθε φορά, πρέπει να υπάρξει μια συνένεση. Και αν δεν υπάρχει συνένεση θα έχουμε σημαντικότατο πρόβλημα. Και ρωτώ την Κομισιόν, σε ποιο βαθμό έχουμε ένα ε, χρονοδιάγραμμα ώστε, εν πάση περιπτώσει, με τους μεγάλους βιομηχανικούς ομίλους να έχουμε μία συνένεση. Γιατί μας ενδιαφέρει και εμάς. Ώστε και εμείς οι πολίτες που είμαστε συνεχώς πιο απαιτητικοί ε, στα θέματα των εκπομπών, γιατί καταναλώνουμε, αγοράζουμε τελικά τα αυτοκίνητα και με αυτό το κριτήριο και στο πλαίσιο των μεταφορών και του τουρισμού θα πρέπει να φτάσουμε σε μια συνένεση. Εάν μείνουμε στα ότι η σύγκριση έμεινε κατά μέρο διότι υπήρχε μια συγκεκριμένη τάση ακαδημαϊκή ή άλλη, θα έχουμε συνεχώς τα ίδια σχόλια και καθόλου επικοδομητικά. Εγώ συμφωνώ με όλες τις ε, τεχνικές και επιστημονικές ε, ε, μελέτες Δηλαδή όταν πλέον βλέπουμε ότι αυτοί που χρησιμοποιούν ποδήλα, ποδήλατο στα αστικά κέντρα τελικά απορροφούν πολύ μεγαλύτερη ποσότητα διοξιδίου από τους άλλους θέλω να πω έχουμε και πρόσθετα προβλήματα και ο κλάδος, είτε μας αρέσει είτε δεν μας αρέσει, έχει μια σημασία, έχει δίνει και θέσεις απασχόλησης, έχει, πρέπει διάφορα και οικονομικά στοιχεία να λάβουμε υπόψη μας. Και νομίζω ότι και η γάμα θα πρέπει, εν πάση περιπτώσει, αυτούς, αυτούς τους κύκλους τους προσαρμογής ε, που θαυμάσια τους έχετε κάνει και σας συγχαίρω, να μην καταλήξουν το κάποιο εργαστήριο κάποιου ε, επιστημονικού Ινστιτούτου να μας πει ότι τελικά όλοι αυτοί οι κύκλοι δεν είναι ε, συγχρονισμένοι μεταξύ τους, δεν μπορούν να συνδυαστούν κτλ. Ε, σας παρακαλώ πραγματικά να επικρατήσει μια συνένεση, να εξευρεθεί μια συνένεση, μια κοινή κατεύθυνση. Είναι πολύ σημαντικό πιστεύω να φτάσουμε σε μια απόφαση που να είναι αποδεκτή και να μπορέσει να εφαρμοστεί. Κάποιοι θα χάσουν λίγο, κάποιοι θα κερδίσουν λίγο, αλλά είναι σημαντικό, εν πάση περιπτώσει, αυτά τα θέματα των, κύκλων που θαυμάσια την για τα έχετε επιτύχει, να μπορέσουμε να τα εφαρμόσουμε σε, σε κάτι που να, που να γίνεται στην πράξη. Σας ευχαριστώ. Thank you very much. Ε, ευχαριστώ πολύ. Ολοκληρώσαμε τον κατάλογο των ομιλητών, ολοκληρώνουμε τον κατάλογο των ομιλητών με τον κύριο Ντάνστ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Υπάρχει συνένεση σχέση με αυτό που πρέπει να κάνουμε και αυτό είναι πολύ ενθαρρυντικό. Ελπίζω ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα ε, σημειώσει όλα ε, αυτά ε, που ακούστηκαν. Ήμουν σε ένα ποτηλιάρισμα πίσω από ένα λεωφορείο που έγραφε Euro 5 από πίσω και υπήρχε ένα πράσινο φύλλο, υπήρχε μια εικόνα ενός πράσινου φύλλου που έβγαινε από την εξάτμιση, το οποίο μου φαίνεται κάπως ε, περίεργο. Ε, το είναι πολύ σημαντικό αυτό. Πάρα πολύ, ο πάρα πολύ καιρό ο κόσμος ακούει ότι τα, οι προδιαγραφές που υπάρχουν αυτή τη στιγμή είναι ε, επαρκής. Δόθηκε προηγουμένως το παράδειγμα του Λονδίνου που θεωρείται μια ε, ζώνη πολύ χαμηλών εκπομπών. Παρόλα αυτά δεν, υπάρχουν, ε, δεν έχουν υλοποιηθεί όλα τα έργα που έχουμε προβλέψει γιατί νομίζαμε ότι τα οχήματά μας ε, πληρούσαν τις απαιτήσει, κάτι που δεν συμβαίνει. Υπάρχει ένα πρόβλημα λοιπόν με την εμπιστοσύνη των πολιτών και αυτό πρέπει να το αποκαταστήσουμε, να μην φτάσουμε στο χαμηλότερο κοινό παρονομαστή, να φτάσουμε στην καλύτερη δυνατή και στην πιο φιλόδοξη ε, κατά το δυνατόν ε, πρόταση, γιατί μόνο μία ευκαιρία έχουμε να τα καταφέρουμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να δώσω τώρα το λόγο στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να απαντήσει. Πάρα πολλές ε, ερωτήσεις ακούστηκαν. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Πρόεδρε και ευχαριστώ για όλα τα σχόλια και τις ερωτήσεις. Θα προσπαθήσω να καλύψω τα περισσότερα από αυτά γιατί κάποια άλλα αφορούσαν τους ε, συντελεστές, ε, αντιστοίχησης, οπότε θα ε, ε, τα αφήσω στο συνάδελφο ε, που θα, που θα καλύψει το θέμα της WLTP. Το ερώτημα ήταν, το ερώτημα που άκουσα, ένα πολύ σημαντικό ερώτημα, είναι γιατί η δική μας Γενική Διεύθυνση είναι η υπεύθυνη. Κοιτάξτε, ε, Ελπίζω ότι δεν θα σας απογοητεύσει η λύση την οποία θα προτείνουμε. Ε, ο λόγος ε, για τον οποίο η δική μας Γενική Διεύθυνση η ανάπτυξη είναι υπεύθυνη είναι γιατί είναι υπεύθυνη για την έγκριση τύπου των οχημάτων ε, Μιλάμε για ε, την έγκριση τύπου εξοπλισμών ε, και με νέο κύκλο δοκιμών που θα μας δώσει τη δυνατότητα να μετρήσουμε σωστά τις εκπομπές αερίων. Γι' αυτό ακριβώς η δική μας Γενική Διεύθυνση, επειδή συνεργαζόμαστε πάρα πολύ με τη Γενική Διεύθυνση Περιβάλλοντος, ε, είναι εδώ δίπλα μου και μάλιστα μου ψηφυρίζουν και απαντήσεις στα ερωτήματα που θέσατε. Πραγματικά έχουμε συγγραμμιστεί στις απόψεις μας και θέλουμε να επιτύχουμε τους ίδιους στόχους. Τώρα, ποιος είναι αυτός ο στόχος, θα σας το πω ε, σαφέστατα. Θέλουμε να υπάρξει πλήρης συμμόρφωση με ε, τα ε, όρια εκπομπών Euro 6. Αυτό θέλουμε να επιτύχουμε με την εργασία μας. Υπήρξαν κάποια σχόλια που αφορούσαν το τι θα προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή όσον αφορά τις ειδικέ τιμές ε, για τους συντελεστές ε, συμβατότητας. Ε, ο τελικός συντελεστής είναι ένα. Και όπως είπα, θα υπάρξει ένα δεύτερο πακέτο RDE ε, σε δύο ε, στάδια και το όριο για το δεύτερο στάδιο είναι ακριβώς αυτό που σας ανέφερα. Το πραγματικό ερώτημα λοιπόν δεν είναι πού θα φτάσουμε, Φυσικά πρέπει να υπάρξουν πολύ σοβαρέ συζητήσει, εντατικέ συζητήσει ε, με τα κράτη-μέλη. Ποιο θα είναι ο ενδιάμεσο συντελεστή. Δεν μπορώ να σα πω αυτή τη στιγμή. Θέλουμε να είναι όσο το δυνατόν χαμηλότερο, αλλά είναι ένα πάρα πολύ περίπλοκο ζήτημα, περίπλοκη διαδικασία και πρέπει να ε, ακούσουμε τι απόψει των κρατών μελών, ε, τι απόψει τρίτων μερών, τη βιομηχανία και πρέπει να υπάρξει ο σωστό συμβιβασμό. Το ερώτημα του κατά θα υπερβούμε αυτό που ζητά η νομοθεσία. Κοιτάξτε, είναι θέμα μεθόδου μέτρησης ε, ε, και διαδικασίας ε, ε των φορητών μετρητών δηλαδή θα, πάρουμε, θα λάβουμε υπόψη μας ε, τους, ε, ε, μετρη, τις μετρήσεις, τις τιμές για το Euro 6 και κάποιο στατιστικό σφάλμα που μπορεί να υπάρχει. Δεν θα αλλάξουμε τα, τις οριακές τιμές, απλώς θα τα συσχετίσουμε με την πραγματικότητα. όσον αφορά τις μελέτες που αναφέρατε, βεβαίως τις γνωρίζουμε, την SST, την TNO και μπορούμε να επιβεβαιώσουμε ότι δυστυχώς ε, οι παραβιάσεις ε, είναι πέντε φορές ε, μεγαλύτερες από αυτές που περιμέναμε να υπάρχουν. Και αυτό πραγματικά πρέπει να το λάβουμε υπόψη μας. Όσον αφορά τις παραβιάσεις, και αυτό είναι μια πολύ ανησυχητική κατάσταση και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι αποφασισμένη να αποκατασταθεί η ομαλότητα, ε, δεν μπορώ να σας πω τι θα γίνει κατά τη διάρκεια των επόμενων μηνών σε σχέση με τις ε, παραδιάσεις των ορίων, αλλά γι' αυτό ακριβώς συζητούμε το πακέτο RDE σήμερα, ε, γι' αυτό ακριβώς θέλουμε να επιμείνουμε στο χρονοδιάγραμμα. Ο στόχος μας, επαναλαμβάνω, είναι να υπάρξει ε, μία πρόταση πριν από το τέλος του έτους, ώστε να αρχίσει να εφαρμόζεται σε δύο στάδια και κατά το 2020 ο συντελεστής συμβατότητας ε, που ορίζει η νομοθεσία να αρχίσει να ισχύει. Νομίζω ότι αυτό, αυτές οι απαντήσεις μου καλύπτουν τις περισσότερες ερωτήσεις σε σχέση με το RDE. Ε, τις δοκιμές σε πραγματικές συνθήκες οδήγησης δηλαδή, ο συνάδελφος θα απαντήσει τα υπόλοιπα, τα ερωτήματα. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Τζοάννα, ε, και ευχαριστώ πάρα πολύ για τα ερωτήματα Κοιτάξτε, πολλοί είπαν ότι δεν θα έπρεπε να, είναι λιγότερο φιλόδοξοι, να καταστούν λιγότερο φιλόδοξοι οι στόχοι. Και αυτό με ενθαρρύνει. Έχουμε τους στόχους διοξιδίου του άνθρακα για, τα 2015, ε, για το 2020. Ε, είναι πολύ συγκεκριμένοι αυτοί οι στόχοι. Αναθεωρήθηκαν πέρυσι και ε, οι συνομοθέτες αποφάσισαν τον Απρίλιο του 2015. Αυτό σας το υπενθυμίζω απλώς. Πρέπει να θυμόμαστε ότι αυτοί ε, οι στόχοι ε, ορίστηκαν βάσει του νέου Ευρωπαϊκού Κύκλου Οδήγησης, του NEDC οι αυτοκινητοβιομήχανοι ε, το έχουν αυτό στο μυαλό τους όταν κατασκευάζουν τα οχήματά τους και με αυτού τους στόχους πρέπει να συμμορφωθούν. Όταν λοιπόν εμείς ερχόμαστε το 2017-2018 και αλλάζουμε αυτό τον κύκλο οδήγησης και πάμε στο WLTP που είναι η παγκόσμια διαδικασία δοκιμών ελαφρών οχημάτων, ε, Ξέρουμε πάρα πολύ ε, καλά τι σημαίνει η αλλαγή αυτή και γι' αυτό ακριβώς υπάρχει αυτή η ιδέα της Συγκρίσιμη αυστηρότητα. Αν έχει κάποιος ένα φορτηγό, ένα αυτοκίνητο το οποίο ε, σχεδιάζεται και πρέπει να ε, ακολουθεί κάποια συγκεκριμένα πρότυπα και να ε, πληρεί κάποιους στόχους, ε, δεν μπορείς μετά να αρχίσει να λες «Α, όχι, ξαφνικά αυτό το όχημα πρέπει να πληρεί και τις προποθέσει του WLTP». Αυτό δεν γίνεται γιατί δεν, δεν είναι συγκρίσιμο κάτι τέτοιο. Γι' αυτό ακριβώς χρειάστηκε να λάβουμε πολύ δύσκολες αποφάσεις ε, της φόρτισης της μπαταρίας, ε, του επίπεδου φόρτισης της μπαταρίας, ε, πίεσης των ελαστικών, όλα αυτά τα πράγματα είναι πτυχές τα οποία, οι οποίες αναπτύχθηκαν εδώ και πάρα πολλές δεκαετίες στο πλαίσιο της NDC. Δεν μπορούμε εν μία νυχτή να τα αλλάξουμε και να πούμε «Α, δεν ισχύουν πια αυτές οι προϋποθέσεις», γιατί ακριβώς δεν ισχύει τότε αυτή η συγκρίσιμη αυστηρότητα που ανέφερα προηγουμένως. Πρέπει λοιπόν να το λάβουμε αυτό και επίση χρειάστηκε να υπάρξει συνένεση με τα κράτη-μέλη, με τι μη κυβερνητικέ οργανώσει, ε, με τη βιομηχανία για το πώ θα εφαρμοστούν όλα αυτά τα πράγματα. Και αυτή τη στιγμή η συνένεση έγκυται στο εξή. Πώ δούλευαν όλα αυτά τα πράγματα στο πλαίσιο του NEDC και πώ θα εφαρμοστούν στο πλαίσιο τη διαδικασία ε, ε, αντιστοίχηση και στο πλαίσιο αυτή τη συγκρίσιμη αυστηρότητας. Ε, και υπάρχει αυτό το θέμα των super credits ε, γιατί γίνεται ο σχεδιασμός βάση ε, του NEDC είτε καλύπτονται από τα 50 χιλιόγραμμα είτε όχι. Καταρχάς δεν έχουμε τη νομική ε, εξουσία να, τα αλλάξουμε αυτό και επίση δεν ισχύει τότε αυτή η συγκρίσιμη αυστηρότητα που ανέφερα. Τα 50 ε, ε, χιλιόγραμμα ελπίζουμε ότι θα συνεχίσουν να ισχύουν στο πλαίσιο WLTP. Δεν είναι μια πρόταση Ευρωπαϊκή Επιτροπής. Αυτή είναι η δουλειά των εμπειρογνωμόνων πριν φτάσουμε στη διαδικασία λήψη αποφάσεων σε πολιτικό επίπεδο. Επίσης, υπήρξε μια πάρα πολύ καλή ερώτηση πότε θα σταματήσει ε, ο συσχετισμός. Αναφέρθηκε το 2025. Ελπίζω νωρίτερα ε, γιατί ε, καταλαβαίνετε δεν θέλουμε ή e να συνεχιστεί αυτή η διαδικασία. Ελπίζουμε κάποια στιγμή το συντομότερο δυνατόν να σταματήσει και αν υπάρχουν ε, κάποιοι στόχοι μετά ε, από το 2020 θα πρέπει οι στόχοι αυτοί να διέπονται από το, τη διαδικασία WLTP. Ένα ακόμη ερώτημα αφορούσε τη χάσμα μεταξύ των δοκιμών στις πραγματικές συνθήκες ε, και ε, την έκθεση TNE. Προφανώς υπάρχει μια διαφορά μεταξύ του κύκλου δοκιμών και της πραγματικής, του πραγματικού κόσμου. Ε, έχουμε και τις δικές μας ε, μελέτες, που επιβεβαιώνουν το μέγεθος του προβλήματος αυτού. Ένας τρόπος να το περιορίσουμε είναι η εισαγωγή του WLTP. Αυτό θα δώσει πιο ρεαλιστική ειδικά νούμερα ε, οδήγησης σε σχέση με το NDC. E θα βασίζεται πάλι σε μέσους όρους. Δεν θα είναι ακριβώς αυτό το οποίο έχει κανείς ως εκπομπές όταν οδηγεί για να πάει σπίτι του. Αλλά ελπίζουμε ότι θα είναι πολύ πιο ε, ρεαλιστικό από αυτό που ε, αναφέρουμε τώρα στους πολίτες μας. Ευχαριστώ. Το Συμβούλιο τώρα. Θέλει να προσθέσει κάτι. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Δεν απευθύνθηκαν σε μένα συγκεκριμένα ερωτήσεις. Δεν θέλω απλώς να υπενθυμίσω, ύστερα από τοποθέτηση του κυρίου Καλχάινς Φλόρεντς, ότι δεν γίνεται διαπραγμάτευση στο Συμβούλιο για τις δοκιμές σε πραγματικές συνθήκες. Η ποιότητα του ατμοσφαιρικού αέρα είναι προτεραιότητα της Λουξεμβουργιανής Προεδρίας. Και σε αυτό εγγράφεται και το ζήτημα της μείωσης των εκπομπών από οχήματα που κινούνται στους δρόμους μας. Παρακολουθούμε λοιπόν την εργασία, αλλά δεν είναι ζήτημα διαπραγμάτευσης απευθείας στο Συμβούλιο. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, λέει ο Πρόεδρος. Μπορούμε να κλείσουμε το θέμα αυτό, ευχαριστώντας την Επιτροπή και το Συμβούλιο για την ευκαιρία να συστήσουμε το θέμα. Επόμενο θέμα στην ημερήσια διάταξη. Στα διάφορα δεν προβλέπει τίποτα προς συζήτηση. Πριν κηρύξουμε το πέρα στη συνεδρία σας, υπενθυμίζω ότι αναμένεται 15 Σεπτεμβρίου να διεξαχθεί η προσοχή μας συνεδρίαση εδώ στις Φρυξέλλες. Ευχαριστώ και καλή σας όρεξη.